Καλημέρα σας. Αύριο να ψηφίσουμε πρώτη την έκθεση Φερχάινεν γιατί θα πρέπει μετά να περάσει σε άλλη επιτροπή για ψηφοφορία. Δεν διαφωνεί κανείς. Εντάξει. Έκθεση Φερχάιν αύριο πρώτο. Πρώτη έκθεση θα, θα τεθεί σε ψηφοφορία. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη έγκριση των πρακτικών από την περασμένη φορά. Αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν ε, ζητήσει κανείς κάποια τροποποίηση, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Θα ήθελα να πω για την ημερήσια διάταξη ότι κάποιες μεταφράσεις δεν υπάρχουν. Βουλγαρικά, τσεχικά, αισθηνωνικά, ε, μαλτέζικα, σουηδικά, πορτογαλικά, σλοβενικά δεν έχουμε. Ολλανδικά μπορεί να μιλάτε, αλλά δεν μεταφράζονται, δεν υπάρχει διερμηνία προς τα Ολλανδικά. Στο φάκελό σας θα βρείτε μια έκθεση για μια ε, για ένα ταξίδι στον Κιμάρες που ήταν πολιτιστική πόλη. Μπορούμε να το διαβάσουμε γιατί μπορούμε να ξαναπάμε εκεί ενδεχομένως για να πάρουμε ε, μια γεύση αυτής της ε, ατμόσφαιρας της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Αύριο θα, ψηφίσουμε, θα ε, να έχετε τις ηλεκτρονικές κάρτες μαζί. Τώρα θα προχωρήσουμε στο σημείο 4. Σημείο 4 λοιπόν και δίνω στον εαυτό μου το λόγο. Τον έχω έτσι κι αλλιώς. Περνάμε στο νέο πρόγραμμα της Κομισιόν για τη διαβίου μάθηση, το πρόγραμμα για εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμό, το πρόγραμμα της Ένωσης. Δεν μιλάμε για πρώτη φορά, γι' αυτό και πέρσι το 2011 το Νοέμβρη υπήρξε πρόταση για τη γενική επαγγελματική κατάρτιση και την ε, νεολαία και τον, τον αθλητισμό, το παρουσίαση η Κομισιόν και θεού θέλοντος από το 2014 θα τρέξει το πρόγραμμα για 7 χρόνια. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων έγινε τέλος Μαΐου και εγώ είχα μιλήσει για κάποια σημεία του προγράμματος, μίλησα και για το όνομά του και για την αρχιτεκτονική του και για την ορατότητα των επιμέρους εκπαιδευτικών τομέων και του τομέα της νεολαίας και τις, ε, τα ελάχιστα ποσά που χρειάζονται για τους τομείς. Εκείνο το κείμενο που είχα παρουσιάσει και πάνω στο οποίο είχα βασιστεί, το έχετε ακόμα. Αυτό έρεται. Ε, απόψε θα πάρετε καινούριο κείμενο με τις νέες παρατηρήσεις μου για τα άλλα μέρη του προγράμματος. Σήμερα θα ήθελα να πω το εξής για το θέμα, για το Erasmus Masters ε, για την γενικότερη διάσταση του προγράμματος και τις γειτονικές χώρες και επίσης θα υπησέλθω σε ορισμένες πτυχές της διαχείρισης του προγράμματος και την πρακτική του υλοποίηση. Επαναλαμβάνω, μιλήσαμε για κάποια θέματα που αφορούσαν τη δομή του προγράμματος. Έχετε σχέδιο. Απόψε θα πάρετε κι άλλο ένα Ίσως το έχετε μπροστά σας ήδη ή θα το πάρετε το βράδυ μέσω διαδικτύου που θα είναι μια περίληψη αυτών που θα σας πω σήμερα. Η Κομισιόν πρόκειται για το Erasmus Masters Guarantee Facility. Η Κομισιόν προτείνει λοιπόν με μια τέτοια διευκόλυνση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια χρηματοπιστωτικά σε τέτοια ε, ιδρύματα θα δίνει μια εγγύηση ότι οι σπουδαστές κάτω από ευνοϊκές συνθήκες θα μπορούν να παίρνουν δάνεια και θα ολοκληρώνουν στο εξωτερικό με αυτόν τον τρόπο τις σπουδές τους στο μάστερ. Αυτό το νέο μέσο στηρίζει την ε, κινητικότητα. Degree Mobility, όπου μπορεί δηλαδή να ολοκληρωθούν οι σπουδές μέχρι το πτυχίο. Και Συμπληρώνονται έτσι τα εθνικά προγράμματα σπουδών που παλιά δεν μπορούσαν να λάβουν χώρα και στο εξωτερικό. Καμιά φορά γινόταν, καμιά φορά δεν γινόταν αυτό. Ελπίζω ότι η νέα ιδέα δεν θα ε, κάνει κάποια κράτη-μέλη να περιορίσουν την δυνατότητα χρηματοδότησης και στο εξωτερικό. Στα στις κανονικές υποτροφίες για μικρότερα χρονικά διαστήματα παραμονής, το Credit Mobility, το ένα ήταν Degree Mobility που είναι ολόκληρο το Master, το Credit Mobility είναι 6 με 12 μήνες. Αυτά τα προγράμματα κινητικότητας Credit παραμένουν και για το Bachelor και για το Master γιατί πολλές φορές μας είπαν ότι τώρα θεωρούν ότι αν το Εράσμους μπορεί να γίνει ολόκληρο στο εξωτερικό, τότε στα πλαίσια του Εράσμους δεν μπορεί κανείς να πάρει credit για τις ε, κανονικές σπουδές. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Το Εράσμους παραμένει για το bachelor και για το master. Όμως υπάρχει κάτι καινούριο, ε, αυτά τα δάνεια δηλαδή για χρηματοδότηση των σπουδών μάστερ. Στο Erasmus Master η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει πάντοτε δάνεια, αλλά κλείνει συμβάσεις η Κομισιόν με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που με τη σειρά τους δίνουν χαμηλότοκα δάνεια, ευνοϊκά δάνεια στους σπουδαστές. Και έχουν και μια εγγύηση ε, που αναλαμβάνει κάποιες ε, ε, δυσκολίες όταν υπάρχουν προβλήματα στην επιστροφή των χρημάτων. 43.000 δάνεια προτείνει η Κομισιόν. Ένα πλήρες δάνειο για ένα χρόνο θα είναι περίπου 12.000 ευρώ και 18.000 ευρώ για δύο χρόνια. Τώρα, για να καλυφθούν οι εγγυήσεις στο διάστημα 2014-2020 που θα είναι περίπου 281 όχι, να καλύψουμε τις εγγύησεις τώρα, από το 2014 με το 2014, 281 ε, εκατομμύρια ευρώ θα βγουν από τον προϋπολογισμό του προγράμματός μας. Αυτό είναι μια ένα λανθάνον ποσό που πρέπει όμως να υφίσταται. Το 2014 το προβλεπόμενο ποσό θα είναι σχετικά μικρό γιατί αρχίζουμε. Θα είναι περίπου 30 εκατομμύρια που θα τα βάλουμε ε, θα τα δεσμεύσουμε και με την ορίμανση του προγράμματος το ετήσιος προϋπολογισμός μέχρι το 2020 θα φτάσει, θα αυξηθεί στα 180 εκατομμύρια. Συμφωνώ ότι τα διάφορα συστήματα επιχορηγήσεων και δανείων παίζουν σημαντικό ρόλο για την κινητικότητα των σπουδαστών. Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα, αλλά ας το συζητήσουμε. Τώρα, στη διάσκεψη του Βερολίνου, στις ε, διαδικασίες της Μπολόνια το 2003, οι Υπουργοί Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι τα κράτη-μέλη τα απαραίτητα, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε οι σπουδαστές, τα δάνεια τα εθνικά και τι επιχορηγήσεις εθνικές να τι χρησιμοποιούν και για το εξωτερικό. Τώρα τα περισσότερα κράτη-μέλη προσφέρουν υποστήριξη για σπουδέ στο εξωτερικό. Όμως οι, οι προποθέσει πρόσβαση είναι διαφορετικές και συχνά είναι απλούστερο να έχει κανείς υποστήριξη για βραχύτερα χρονικά διαστήματα σπουδών στο εξωτερικό από ότι να καλυφθεί το διάστημα όλων των σπουδών. Είμαι υπέρ τη ιδέας, κινητικότητα όχι μόνο για βραχύτερα χρονικά διαστήματα σπουδών, αλλά για ολόκληρε τι σπουδέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Erasmus Masters όμω θα πρέπει να προετοιμαστεί πάρα πολύ προσεκτικά, να δοκιμαστεί και δεν θα πρέπει να πάρουμε ε, πίσω τα κίνητρα από τα κράτη-μέλη ε, ώστε να βελτιώνουν τα υφιστάμενα εθνικά του συστήματα περαιτέρω. Ε, που χρειάζονται διευκρινήσεις. Στα εξή σημεία στο Erasmus Masters. Πρώτον, η πρόταση της Κομισιόν δεν ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με τις απώλειες λόγω των δανείων που θα ε, προκύψουν ενδεχομένως στο δεύτερο μισό του προγράμματος όταν θα είναι προς το τέλος του το πρόγραμμα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το πώς το Erasmus Masters θα εφαρμοστεί σε τελευταία ανάλυση. Πρέπει να ξέρουμε πόσο συντονισμός και διοίκηση, διαχείριση χρειάζονται για το νέο σύστημα. Τρίτον, δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου για να, εξασφαλίζουμε ότι οι σπουδαστές θα προχωρούν στις σπουδές τους και πράγματι θα ολοκληρώνουν τις σπουδές. Είναι πολλά τα ερωτήματα που σημειώνω. Ελπίζω να με ακούνε και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν. Α, ωραία. Τέταρτον, με βάση την πρόταση της Κομισιόν, οι σπουδές σε κάθε χώρα που συμμετέχει θα μπορούν να συνάπτουν δάνειο ανεξάρτητα από το που ζουν την εποχή εκείνη ή που θέλουν να σπουδάσουν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει εδώ να ε, ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα ούτως ώστε οι σπουδαστές πρωτίστως να είναι σε κάποια σημαντική χώρα για αυτούς, είτε στη χώρα διαμονής τους ή στη χώρα που θέλουν να σπουδάσουν. Από εκεί δηλαδή να ζητούν να πάρουν το δάνειο. Αυτό είναι για το Erasmus Masters. Τώρα, περνάω στο, στη διεθνή διάσταση του προγράμματος που έχει συζητηθεί πολύ. Το νέο πρόγραμμα δεν προωθεί μόνο την κινητικότητα μεταξύ των ε, συμμετεχουσών χωρών, αλλά μεταξύ συμμετεχουσών, συμμετεχουσών χωρών και τρίτων χωρών, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά μεταξύ ημών και τρίτων χωρών επίσης. Η πρόταση της Κομισιόν, όλα τα προγράμματα, τα εντάσσει εδώ στο Erasmus Mundus όπως και, και λειτουργεί όπως και άλλα διμερεί προγράμματα. Ε, εγώ είμαι υπέρ αυτής της απλουστευμένης αρχιτεκτονικής για την διεθνή διάσταση στον τομέα της παιδείας. Βρίσκω ότι είναι καλή. Για την κινητικότητα από τρίτες χώρες και για τη διεθνή συνεργασία θα διατεθούν κονδύλια από πέντε εξωτερικά μέσα. Είναι το μέσο για την αναπτυξιακή συνεργασία, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας, το μέσο της βοήθειας προσέγγισης, το εκείνο για την εταιρική σχέση και τέλος το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Συνολικά για την διεθνή διάσταση του προγράμματος προβλέπονται 1,8 δις είναι το 2% ολόκληρου του προϋπολογισμού για όλα τα εξωτερικά αυτά μέσα. Για την χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων θα ισχύουν οι κανόνες του νέου προγράμματος. Τονίζω εδώ ότι οι αρχές, οι στόχοι και οι προτεραιότητες αυτών των εξωτερικών μέσων θα πρέπει να ε, την χάνουν σεβασμού. Τώρα για το μέσο για την αναπτυξιακή συνεργασία χρειάζεται προσοχή γιατί μόνο η κινητικότητα των σπουδαστών από τρίτες χώρες σε συμμετέχουσες χώρες θα υποστηρίζεται. Δεν θα είναι δυνατόν σπουδαστές από την Ευρώπη να πάνε σε τρίτες χώρες με αυτό το πρόγραμμα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να χρηματοδοτούνται από κονδύλια αναπτυξιακά. Αυτό έχει να κάνει με τα αυστηρά κριτήρια που ισχύουν για το συγκεκριμένο μηχανισμέσο. Ότι δηλαδή θα πρέπει η ανάπτυξη σε εκείνες τις χώρες να προαχθεί και όχι να βοηθήσει τους σπουδαστές τους δικούς μας να πάνε εκεί. Η διεθνής διάσταση του τομέα της παιδείας θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη διάρκεια των προγραμμάτων, του, του προγράμματος που είναι 7 ετής, θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποια ευελιξία, ούτω ώστε η διεθνή κινητικότητα να λαμβάνει υπόψη και να περιλαμβάνει επίσης και την επαγγελματική κατάρτιση, ούτω ώστε η ανάπτυξη αυτού του κομματιού να υποστηριχθεί και σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα γειτονικές χώρες. Προχωρώ στο ρόλο των ε, χωρών των γειτονικών. Το Συμβούλιο, στο γενικό προσανατολισμό του, ε, έδωσε τη δυνατότητα στις γειτονικές χώρες να γίνουν συμμετέχουσες χώρες αν έχουν διμέρει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή, αυτό σημαίνει ότι όλες τις δυνατότητες αλλά και όλες τις υποχρεώσεις θα τις έχουν όπως ακριβώς και οι συμμετέχουσες χώρες. Ε, αυτό έχει πρακτικές συνέπειες. Πρώτον, για να συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα, οι χώρες αυτές θα πρέπει αφενός να ε, δημιουργήσουν ε, μια εθνική υπηρεσία, δεύτερον θα πρέπει να πληρώσουν μια κάρτα εισόδου το αν θα επιστρέφονται οι δαπάνες αυτές δεν μου είναι ξεκάθαρο, δεν μου είναι γνωστό. Ενώ κονδύλια από το μέσο γειτονία, αν δεν υπάρχουν ε, δεν, θα δεν θα είναι πια αν γίνουν συμμετέχουσες χώρες ε, ε, δεν θα είναι γειτονικέ, δηλαδή αν καλύπτονται από το καθεστώς που διέπει τις συμμετέχουσες χώρες ε, θα χρηματοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο και δεν θα παίρνουν πια λεφτά από το μέσο γειτονία. Επίσης και για ε, κεντρικές ε, εκδηλώσεις θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον, όπως ας πούμε οι συμμαχίες της γνώσης κλπ. Θα μπορούν να συμμετέχουν και στις αποκεντρωμένες δραστηριότητες όπως κινητικότητα, συνεργασία με ε, ιδρύματα ε, εταίρους αν, το επαναλαμβάνω, έχουν κάνει ε, μια διμερή διευθέτηση με άλλες χώρες. Εγώ υποστηρίζω το πρόγραμμα αυτό, ναι, ε, να ανοίξει και να υπάρξει δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του προγράμματος. Όμως δεν πρέπει να ε, αρνηθούμε το γεγονός ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τις τρίτες χώρες τι σημαίνει αυτό από άποψη δαπανών για αυτές. Και θα πρέπει βέβαια να είναι σε θέση να υπομισθούν αυτές τις δαπάνες. Είναι δηλαδή πράγματα από αυτά που πρέπει να τα έχουμε πολύ ε, στο μυαλό μας. Και περνώ τώρα σε ένα άλλο ωραίο σημείο. Ε, εκτελεστικές και κατεξουσιοδότηση πράξης. implementing και delegated. Με βάση της πρότασης της Κομισιόν, μιλάτε, ε, έχουμε ένα ετήσιο πλάνο, το οποίο με εκτελεστικές ε, πράξεις θα αποφασίζεται. Εκεί εμείς δεν έχουμε συμμετοχή. Στα ετήσια προγράμματα εργασίας θα πρέπει να υπά, περιγράφονται οι στόχοι, οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν και μια ενσωμάτωση ε, στον προϋπολογισμό. Και μετά θα ε, χρησιμοποιούνται και κριτήρια αξιολόγησης και θα υπάρχει επίσης και το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης. Υπενθυμίζω ότι με βάση το άρθρο 290 της συνθήκης τα στοιχεία που μπορούν να καλύπτονται και να αποφασίζονται από εκτελεστικές πράξεις είναι αυτά τα οποία αφορούν την διεξαγωγή του μελλοντικού προγράμματος πολλά από τα θέματα που προανέφερα, όπως οι στόχοι, τα κριτήρια αξιολόγησης, δεν αφορούν μόνο τη διεξαγωγή του προγράμματος, την υλοποίησή του, αλλά στόχο έχουν να συμπληρώσουν ορισμένες διατάξεις ή και να τις τροποποιήσουν. Γι' αυτό με εξουσιοδότηση πράξης ε, θα πρέπει να αποφασίζονται τα θέματα αυτά βάσει του άρθρου 291 της συνθήκης, πράγμα που ε, ισχύει και για το Creative Europe, τη Δημιουργική Ευρώπη. Τα ίδια συζητούνται και εκεί. Προχωρώ στους δείκτες ε, για την αξιολόγηση του προγράμματος. Η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει για κάθε στόχο δείκτες για την παρακολούθηση, monitoring και την μετέπειτα αξιολόγηση του προγράμματος. Εγώ την ιδέα αυτή την υποστηρίζω. Οι δείκτες θα πρέπει να υπάρχουν στο βασικό δίκαιο, ούτω ώστε να ισχύουν και να εφαρμόζονται από την αρχή του προγράμματος. Και για τη συνοχή του κειμένου θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα σε ένα παράρτημα. Έτσι λέμε εμείς. Το νομικό του καθεστώς δεν επηρεάζεται έτσι, γιατί τα ε, ε, αυτά τα παραρτήματα, είναι κομμάτι του προγράμματος. Τώρα, ε, με τη νέα ε, ορθολογική αρχιτεκτονική του προγράμματος, η Κομισιόν προτείνει να υπάρξει μία μόνο επιτροπή του προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, το, προ... το νέο πρόγραμμα δεν καλύπτει μόνο διαφορετικούς τομείς παιδείας όμως, όπως διεθνή συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά ε, επεκτείνεται και στην νεολαία και τον αθλητισμό. Και αυτή η ετερογένεια μπορεί να ληφθεί υπόψη αν η επιτροπή του προγράμματος ε, διαβουλεύεται με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά ανάλογα με το θέμα το οποίο θα πραγματεύεται. Οι εθνικές αρχές λοιπόν και οι υπηρεσίες, εμείς προτείναμε αυτό να τεθεί στα πλαίσια της επικουρικότητας και κάθε χώρα να αποφασίζει ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για τη διαχείριση του προγράμματος. Οι μικρότερες χώρες θα έχουν μία υπηρεσία, η Γερμανία θα έχει περισσότερες υπηρεσίες. Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα όμως και πήγε καλά. Όμως να είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να δοθούν περισσότερα χρήματα για τη διαχείριση του προγράμματος. Ο αριθμός των ε, υπηρεσιών θα αποφασίζεται από τα κράτη-μέλη. Και αυτό το τελευταίο βρίσκει σύμφωνο και το Συμβούλιο και η Προεδρία με την οποία είχα μια πολύ ωραία συζήτηση και μπορούσα μάλιστα να ε, συνεννοηθώ στα γερμανικά. Εντυπωσιάστηκα, συνεννοήθηκα πάρα πολύ ωραία στα γερμανικά με την Κυπριακή Προεδρία. Ε, λοιπόν, σταματώ εδώ. Δεν επανέλαβα αυτά που είχα πει την περασμένη φορά. Δεν θα ξαναρχίσουμε εκ του μηδενός. Τα έχετε αυτά γραπτός. Παρακαλώ τώρα αυτά που δεν καταλάβατε, α, τις παρατηρήσεις που θέλετε να υποβάλλετε, τώρα είναι η ώρα να τις υποβάλλετε. Για τις ε, λεπτομέρειες, για τα περιεχόμενα, για τους στόχους, δεν θα μιλήσουμε τώρα. Αυτό θα το κάνουμε το Σεπτέμβριο όταν θα υποβάλω και εγώ την έκθεσή μου. Όλες τις ιδέες που έχετε για το πώς θα βελτιωθεί το περιεχόμενο του Εράσιμους ή του Κομένιου ή δεν ξέρω τι άλλο, αυτά θα γίνουν το Σεπτέμβριο αφού θα έχετε δει ε, καθ' την πρότασή μου. Σε αυτό το σημείο αυτά ήθελα να ξεκαθαρίσω, διότι το κείμενο σύντομα θα πάει για μετάφραση. Λοιπόν, για να δω μήπως ξέχασα κάτι. Δεν μίλησα για τον αθλητισμό, δεν χρειάζεται τώρα να το κάνουμε αυτό. Για την νεολαία, είπαμε ότι θα έχουμε ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό για την νεολαία ο συνάδελφος Λούκα δεν είναι εδώ. Ε, στην πρότασή του δεν έχει προβλέψει ειδική γραμμή για την ε, νεολαία, ε, αλλά, την νεότητα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Αν συμπεριληφθεί πρέπει να υπάρχει κεφάλαιο με ειδική γραμμή του προϋπολογισμού. Κλείνω λοιπόν τις παρατηρήσεις μου. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Και σας δίνω το λόγο. Κυρία Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μιλήσω αγγλικά, μια και δεν υπάρχει σλοβαγική διερμηνία και δεν φαντάζομαι ότι κανείς ξέρει τη γλώσσα μου άλλος. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω με, την, ε, με, το, με τη διευκόλυνση για την πίστοση ε, για, τους, για τις σπουδές. Ε, λοιπόν, αυτές οι υποτροφίες οι οποίες υπάρχουν ήδη λειτουργούν πάρα πολύ καλά και επομένως στο μέλλον καλό θα είναι να ενδυναμωθούν και με άλλου είδους δάνεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτήν την Grand Facility και να συνεχίσουμε και με τα δάνεια. Επίσης θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι όλα όσα αποφασίσει το Κοινοβούλιο θα είναι καλά για τους ε, φοιτητές. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θεωρούν, φοβούνται μάλλον, ότι αυτές οι νέες διευκολύνσεις θα αντικαταστήσουν τις παλές, οι οποίες όμως λειτουργούν πολύ καλά. Ε, έχοντας συζητήσει με πολύ κόσμο, έχοντας συζητήσει και με τους ενδιαφερόμενους, με τους φοιτητές δηλαδή, διαπιστώνομαι ότι όλοι θέλουν την εξέλιξη, όχι όμως την αντικατάσταση. Επίσης θα πρέπει να ακολουθηθεί η προϋπόθεση ότι αυτά τα δάνεια θα έχουν καλές συνθήκες όσον αφορά την αποπληρωμή τους ας πούμε, η οποία θα πρέπει κατά την άποψή μου να ξεκινήσει αφού αρχίσουν οι φοιτητές να έχουν εισόδημα, αφού θα έχουν δηλαδή βρει ε, κάποια θέση απασχόλησης για αμέσως μόλις τελειώσουν ε, τη σχολή. και με αυτόν τον τρόπο θα δεχτούν αυτά τα δάνεια οι φοιτητέ. Έχω και άλλα να πω, αλλά δεν θέλω να μιλήσω με πολλή λεπτομέρεια. Ένα άλλο σημείο τώρα, όσον αφορά τον προπολογισμό. Η πρόταση ενό ποσοστού της 100 είναι κατανοητό. Μπορώ να συμφωνήσω, όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε και το ποσοστό της 100 ανατμήμα. Ε, θα πρέπει να υπάρχει σχετική ευελιξία Καταλαβαίνω βεβαίω αυτό που λέτε, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να βρεθεί, να υπάρξει κάποια ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος, ε, στην οποία θα πρέπει βεβαίως να εμπλακεί και το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε ε, εάν ε, πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά τη δομή, τη διάρθρωση, την κατανομή, σίγουρα στην ενδιάμεση αξιολόγηση να συμμετέχει το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει και σε διάφορες τροποποίησεις. Κάτι άλλο σημαντικό ε, για τα grants και για την κινητικότητα ε, κατά την άποψή μου είναι σοβαρό κυρίως για χώρες οι οποίες ε, έχουν χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο ας πούμε από τη χώρα μου είναι δύσκολο να φύγουν οι φοιτητές και να ζήσουν σε άλλες χώρες ακολουθώντας και προγράμματα ανταλλαγών τύπου Εράσμους κλπ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά και το ποσό το οποίο δίνεται στους φοιτητές, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο βιωτικό επίπεδο της χώρας από την οποία προέρχεται ο φοιτητής, αλλά ε, και το βιωτικό επίπεδο ε, της χώρας στην οποία θα ζήσει ο φοιτητής. Δεν είχα τελειώσει, δεν είχα τελειώσει. Ήθελα απλώς να πιω λίγο νερό. Sorry, sorry. Okay, I will I will be fast. Uh, then on uh, the mobility of the secondary education, I agree with. Όσον αφορά τώρα την κινητικότητα, συμφωνώ δηλαδή ότι θα πρέπει ε, να ε, ξεκινήσει αυτή η κινητικότητα όσο γίνεται γρηγορότερα και εν πάση περιπτώσει αν τα δεχτούμε έτσι όπως τα είπατε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο Erasmus Mundus. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, πριν από μερικές εβδομάδες ε, συμμετείχα σε ε, συζήτηση που είχε οργανώσει η Ένωση του Erasmus Mundus και υποσχέθηκα στους ενδιαφερόμενους ότι θα, θα κρατηθεί αυτό, θα διατηρηθεί το όνομα αυτό. Είπες πολλές φορές, Ντόρι, ότι μας πήρε καιρό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία θα πρέπει να τα καταλάβουν πρώτα. Ε, οι πολίτες ήδη πριν αρχίσουν να συμμετάσχουν. Ε, επομένως ήταν δύσκολο να γίνει ορατή αυτή η δυνατότητα. Τώρα, τώρα που έγινε γνωστό το όνομα, αν αλλάξει ε, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Ε, είναι δύσκολο λοιπόν να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Εάν αρχίσουμε το όνομα του προγράμματος ε, δεν θα καταλάβουν ούτε το γιατί ε, και θα μπερδευτούν οπωσδήποτε. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό ναι είναι για τους πολίτες της Ευρώπης αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για όλους τους Ευρωπαίους. Αν θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας, ε, τις αρχές μας, ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε και κάποια ονόματα και κάποιες αρχές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και μία συνέχεια. Αυτά ήθελα να πω. Πολύ καλή δουλειά, θα σας στηρίζω και να τη συνεχίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Ε, η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν έχω να ε, προσθέσω πολλά. Αλλά λίγα. Μπορούμε να πούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν υπογραμμίζει πολύ τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα μπορούσε να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και στον επαγγελματικό τομέα η κινητικότητα των σπουδαστών και να επεκταθεί και σε πιο ελεύθερες δραστηριότητες στον τομέα της παιδείας. Για τις τρίτες χώρες οι δυνατότητες περιορίζονται στα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά καθόλου, δεν υπάρχει καθόλου κινητικότητα στη γενικότερη εκπαίδευση. Θα ήταν σημαντικό στη συνεργασία με τις τρίτες χώρες να συμπεριλάβουμε και την επαγγελματική κατάρτιση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η κινητικότητα όπως και στο Κομένιους. Τώρα, Δύο λόγια για τα δάνεια, τα εγγυημένα δάνεια. Ίσως η Κομισιόν δεν αξιολόγησε ακριβώς τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην προσφορά ε, από πλευράς κρατών μελών στον τομέα της παιδείας και πώς ε, θα συντονιστούν με τα εθνικά συστήματα. Εδώ χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες, αξιολόγηση και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα δανείων ε, στην κινητικότητα. Αυτοί που ολοκλήρωσαν τις σπουδέ τους ε, θα μπορούσαν να... Ίσως δυσκολεύονται αν έχουν πάρει για παράδειγμα δάνειο σε χώρα με ε, υψηλό κόστος ζωής και επιστρέψουν στην πατρίδα τους, μπορεί να έχουν πρόβλημα να επιστρέψουν το δάνειο. Θα είναι πιο δύσκολο για εκείνους από ό,τι για άλλους. Ε, επίσης στον αθλητισμό υπάρχει για πρώτη φορά και εδώ ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για τον αθλητισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ιστορική η πρόταση αυτή και γι' αυτό πρέπει να την υποστηρίξουμε και να την προωθήσουμε, αν και χρειάζονται βέβαια συγκεκριμένα μέτρα εδώ, γιατί η πολιτική δεν είναι αξιόπιστη αν δεν συμπεριλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα. Ε, ε, η οικονομική εποχή τώρα είναι δυσχερής, αλλά παρόλα αυτά καλό είναι να υποστηρίξουμε τον αθλητισμό και εμείς ως Κοινοβούλιο. Ε, η παρουσίασή σας ήταν εξαιρετική. Όπως σας είπα δεν είχα να προσθέσω πολλά, απλώς κάποιες παρατηρήσεις και προς την ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ η Πέτρα Κάμαφέφερ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις κάτι που μου φαίνεται σημαντικό και συμφωνώ και με την Κατερίνα Νεβεντάλοβα για, τις, ε, για τον ε, ε, τρόπο υλοποίησης. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσουν τα, οι, οι, οι πρακτικές συνθήκες επιστροφής των δανείων κλπ. Επίσης, τι θα γίνει με τις εγγυήσεις που δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί δεσμεύουμε αρκετά σημαντικά κονδύλια, ούτω ώστε να εγγυηθούμε για δάνεια που ίσως δεν θα επιστραφούν. Ελπίζομαι ότι δεν θα χρειαστούν αυτά τα κονδύλια γιατί θα επιστραφούν τα δάνεια. Αλλά τι θα γίνει, τα κονδύλια αυτά που θα είναι η εγγύηση θα παραμείνουν στον προϋπολογισμό μας και μπορούν, θα μπορούν στο τέλος του χρόνου αυτά τα χρησιμοποίητα να πάνε για άλλους σκοπούς. Θα μπορούν να μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο και πώς θα, θα επιστρέφουν στα κράτη-μέλη, ίσως και πώς. Μιλάμε για 281 εκατομμύρια ε, καθ' όλο το διάστημα, τη διάρκεια του προγράμματος. Είναι πολλά χρήματα. Θα μπορούσαμε κάποια να τα χρησιμοποιήσουμε πολύ καλά σε άλλες πτυχές του προγράμματος. Καλό είναι λοιπόν να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ε, στην, επίσης, ε, το credit mobility για αυτούς που ε, παρακολουθούν το μάστερ. Υπήρξαν κάποιες ε, αντιρρήσεις για το αν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα και το μάστερ. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι διατυπωμένο ξεκάθαρα ε, το θέμα. Ίσως η Κομισιόν να το ήθελε να το προβλέψει, δηλαδή ότι και τα δύο θα ισχύουν, δηλαδή και το καινούργιο και το παλιό σύστημα να τους καλύπτει. Αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της διαφάνειας στη νομική γλώσσα για να ξέρουν όλοι τι ακριβώς εννοούμε. Ας δούμε λοιπόν μήπως μπορεί να βρεθεί μια σαφέστερη διατύπωση για να μην υπάρχει, να μην επιδέχεται καμία παρερμηνία το θέμα. Ευχαριστώ πολύ θα πω κι εγώ κάτι ε, πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν και στον επόμενο μιλτή. Για το αυτό που είπες τελευταία, Πέτρα, το τόνισα ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ε, degree mobility και credit mobility. Η credit mobility είναι δυνατή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών. Η degree mobility είναι αυτό το οποίο εννοούμε ε, με το μάστερ, στη διάρκεια του μάστερ. Εκεί χορηγείται. Αν όμως δεν το θέλεις για δύο χρόνια, αν θέλεις να πας στο εξωτερικό για έξι μήνες στα πλαίσια του μάστερ, μπορεί να γίνεις στα πλαίσια του credit mobility. Αυτό το λέει καθαρά και το είπα και εγώ το. Δεύτερον, έχεις δίκιο με τις εγγυήσεις που ρωτάς τι θα τα κάνουμε τα χρήματα που θα υπάρχουν. Το 2014 δεν θα χρειάζεται τίποτα, το 2015, το 2016 ίσως χρειαστεί κάτι. Πάμε στο 2017. Στο τέλος του προγράμματος θα έχουν μαζευτεί πολλά χρήματα και το ερώτημα είναι θα τα κρατήσουμε όλα ούτω ώστε να χρηματοδοτήσουμε κάποια πράγματα. Εδώ θέλουμε την απάντηση της Κομισιόν. Κύριε Κορέλ, ίσως ε, μπορείτε να μας πείτε. Τώρα, οι τρόποι επιστροφής των χρημάτων, των δανείων, και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ε, τώρα, η Credit Mobility και η Degree Mobility. Δεν είναι παλιό και καινούριο πρόγραμμα. Το ένα παραμένει, το άλλο προστίθεται. Για τον αθλητισμό, Χάνο. Δεν μίλησα για τον αθλητισμό, γιατί είχα μιλήσει την περασμένη φορά. Νομίζω ότι ε, χαιρόμαστε που έχουμε αυτά, έστω και αυτά τα λίγα ε, θέλουμε βέβαια το μαζικό αθλητισμό κυρίως να υποστηρίξουμε και την συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς κλπ. Αυτά θέλαμε να πετύχουμε και θέλαμε και ε, εταιρικέ σχέσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρόσθετη χρηματοδότηση. Να σας πω όμως και κάτι ακόμα που το ξέχασα πιο πριν. Ψάχνοντας τα προβλήματα παρατήρησα ότι τελευταία ε, συνέβη κάτι που δεν ήταν ωραίο. Δηλαδή η Κομισιόν ξαφνικά τον ΦΠΑ τον ζήτησε πίσω. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένα πρόγραμμα, ας πούμε, ε, οι άνθρωποι μάζευαν τις αποδείξεις, τις των ταξί και όπου υπήρχε ΦΠΑ έπρεπε να αφαιρεθεί και να επιστραφεί θα λέγαμε. Εν τω μεταξύ άλλαξαν τα πράγματα γιατί είδε η Κομισιόν ότι δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα και το άλλαξε. Όμως θα ήθελα με κάθε σαφήνεια να πω ότι ΦΠΑ δεν υπολογίζεται και σε αυτά που πληρώνουμε εδώ. Η οικονομική βοήθεια για κινητικότητα πρέπει να, να... να μην περιλαμβάνει ΦΠΑ. Ε, ούτε κοινωνικές ε, εισφορές. Και αυτό ισχύει και για τα ιδρύματα τα ενδιάμεσα, γιατί δεν παίρνει ο καθένας άμεσα τα χρήματα απευθεία, ε, μπορεί να το πάρει και μέσω κάποιων τοπικών φορέων ενδιάμεσων. Άρα λοιπόν, ούτε στο πρόγραμμά μας δεν μπορούμε να το γράψουμε αυτό, γιατί υπόκειται στην επικουρικότητα. Αλλά επειδή η Κυπριακή κυβέρνηση παρίσταται ε, με ξέχοντες εκπροσώπους θα ήθελα να πω ότι ίσως στο Συμβούλιο θα, θα, θα μπορούσε να τονίσει ότι αυτά που δίνουμε δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, σε εφορολογία και σε κοινωνική, κοινωνικές εισφορές. Δεν είναι δυνατόν το κράτος να ωφεληθεί από αυτά τα οποία ε, έφτασαν στα κοινοτικά ε, ταμεία δεν μπορούμε να τα ζητήσουμε, είναι η επικουρικότητα. Αλλά το Συμβούλιο θα πρέπει να το δει προσεκτικά αυτό, γιατί υπήρξαν και πολλές καταγγελίες πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, άκουσα ορισμένες ερωτήσεις, ακούσαμε ερωτήσεις που μου φαίνεται ότι ήρθε η ώρα ο κύριος Κορέλ να τις απαντήσει. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κυρία Συγκεντρία. Σας ευχαριστώ όλους και όλες εδώ έχουμε μια σειρά ερωτήσεων, να προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Και αν δεν καταφέρω θα ξαναπροσπαθήσω. Πρώτα πρώτα. Όσον αφορά την κινητικότητα, καλά τα λέτε. Ακριβώς σύμφωνα με την ε, κυρία Νελάτοβα, όσον αφορά την συμπληρωματικότητα μεταξύ δανείων και υποτροφιών. Το είπατε κι εσείς. Εδώ μιλούμε για την κινητικότητα των πιστώσεων, μιλούμε για δάνεια, και δεν θα πρέπει επομένω το ένα να βοηθά το άλλο. Τώρα, κάποιες ε, ερωτήσεις που αφορούν το έγγραφο, άλλες που ανέφεραν οι αγορητές. Η πρώτη αφορά το τι συμβαίνει με, τα, με τους πόρους που καλύπτουν αυτή την εγγύηση. Μένουν τα χρήματα εκεί, αυτή είναι η απάντηση. Γιατί ο τρόπος διαχείρισης που προβλέπετε είναι μέσα στο EIF και ούτω καθεξής. Οπότε βεβαίω ο κύκλος ζωής των δανείων θα είναι μεγαλύτερος από κοινών του προγράμματος. Ένα, δύο έτη μελετών, διακοπές που θα περιληφθούν εκεί και κατόπιν θα έχουμε κάποιο μακρόπνοη ρύθμιση αποπληρωμής. 15-20 χρόνια δηλαδή. Άρα τα χρήματα είναι εκεί, ούτω ώστε να μπορέσει κανείς να στηρίξει την εγγύηση. Τώρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, τι προβλέπετε. Ότι χρήματα αποδεσμεύονται από αυτή την υποχρέωση να καλύπτεται η εγγύηση, θα γερνούν στο δανείο του μέσου, του χρηματοδοτικού μέσου. Αυτά συμφώνησαν τα τρία δεσμικά όργανα στα πλαίσια του Δημοσιονομικού Οργανισμού. πάντως είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι τα χρήματα πρόκειται να διαβαστούν το ΕΕΦ, θα χρησιμοποιηθούν ω εγγύηση και μια που τα δάνεια θα είναι πιο μακρόβια, θα πρέπει να υπάρχουν ε, αυτά τα χρήματα, τότε δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση για τα χορηγούμενα δάνεια. Τώρα, στον αφορά νέο μηχανισμό συντονισμού. Όπως γνωρίζετε, Πρόεδρε, είχαμε τη μελέτη βιωσιμότητας και δίναμε όλα τα συμπράσματα πλην ενός. Τι έλεγε αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να διαχειριστεί το σύστημα και λέμε όχι αυτό δεν δημιουργήσει γραφειοκρατία και διοικητικές δαπάνες. Επομένως, το EAF, το οποίο έχει εμπειρία, θα κάνει τη διαχείριση και θα έχουμε μετά τους διαφόρους ενδιαμέσους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν ασκείται έλεγχος. Βεβαίως και ασκείται πρώτα πρώτα πριν δοθεί το δάνειο, τέλος πάντων έτσι ο οικονομικός ε, ενδιάμεσος θα πρέπει να διαπιστώσει ότι ο φοιτητής ε, κάνει μεταπτυχιακά μάστερ σε κάποια διαφορετική χώρα του, από την χώρα κατοικίας και επίσης αν έχουμε ετή περίοδο για το δάνειο, γιατί έχουν πολλά μάστερ διετή, τότε η δεύτερη δόση δεν πρόκειται να εκταμιευθεί εάν δεν υπάρξει επιτυχία για το πρώτο έτος για να εξαρτηθεί ότι όντως σπουδάζει ο φοιτητής. Μισό λεπτό διακοπή του κύριε Ποιος ασκεί τον έλεγχο. Ότι πραγματικά ο φοιτητή σπουδάζει, ο οικονομικός ενδιάμεσος, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εκείνοι έχουν αναλάβει τον κίνδυνο. Θα πρέπει για ένα υψηλότερο κίνδυνο να δώσουν περισσότερα χρήματα αν δεν τα καταφέρει την πρώτη χρονιά. Άλλο σημαντικό το οποίο είπατε όλοι. Το θέμα της ισότητας των όρων χωρίς δανεισμό. Ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το δανεισμό. Πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Εξασφαλίσουμε ναι. ότι θα υπάρχει. Και η μόνη εγγύηση που θα πρέπει να απαιτεί ο χορηγόν το δάνειο είναι απόδειξη ότι έχει εγγραφεί σε μαθήματα για μάστερ ο ετών το δάνειο. Τώρα, το άλλο μπορεί να φερθεί, δηλαδή γιατί είναι αντικειμενικό, θα πρέπει να είναι με όρους ισότητος, θα πρέπει να μην ξέρει κανέναν κοινωνικά και θα πρέπει να είναι ελκυστικό στους φοιτητές αλλά και στους οικονομικούς παράγοντες. Αλλιώς κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Αλλά θα πρέπει να ξεχαστεί το ότι όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σε διακοπέ. διακοπές, ε, ε, να είναι δίκαιοι οι όροι, αλλά να είναι και αρκετά ελκυστική ούτως ώστε να συμμετάσχουν οι, αυτοί οι οικονομικοί ενδιάμεσοι δάλους, κανείς δεν θα θέλει να συμμετάσχει. Θα πρέπει όμως να αναδύονται ξεκάθαρα οι σκοποί κάθε φορά. Όσον αφορά τη συμβατότητα μεταξύ των αυτών των δανείων και των εθνικών δανείων. Είπαμε ότι να είναι απολύτω συμβατά. Μια από τα εθνικά δανεία που έχουμε προσπαθούν είναι ικανοποιητικά, όμω υπάρχει ένα κενό όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο. εδώ μπαίνει ο ρόλο τη πρότασή μα για τη συμπληρωματικότητα άλλο τον κύριο Πακ για το χώρο στον οποίο θα, απευθύνονται ότι για τη χορήγηση οι φοιτητέ Εδώ πρέπει να προσέξουμε. Προσοχή να τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Να μην υπάρχει διάκριση επί τη βάση φίλου, εθνικότητος, αλλά να υπάρχει κάποια σχέση με το ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο, έστω μπορεί να είναι ε, τόπος κατοικίας ή δανείο. Για τη συμπληρωματικότητα τώρα δανείων και υποτροφιών, εδώ έχουμε σαν σημαντικό παράγοντα το επίπεδο των δανείων. Αυτό πρέπει να εξεταστεί στο σοβαρά. Και σήμερα, όταν μιλούμε για το κόστος διαβίωσης, εννοούμε τη χώρα όπου θα γίνουν σπουδέ, όχι τη χώρα προελεύσεως. Επομένως αυτό θα πρέπει να είναι διορθωτικός συντελεστή. Για να καλύψει αυτούς που έρχονται από χώρα όπου είναι κατώτερο το δυτικό επίπεδο από τη χώρα των σπουδών. Ένα άλλο γενικό θέμα, το οποίο αναφέρθηκε, είναι η ανωτάτη παιδεία σε σχέση με άλλους τομείς. Το ξανασυζητήσαμε. Νομίζω όμως ότι σαφώς αυτό το πρόγραμμα θέλει συνολικά να καλύψει όλους τους τομείς. Και τις ε, τυπικές, παραδοσιακές και τις μη παραδοσιακές μορφές. Πάμε για κοινά μάστερ. Ε, φυσικά, εκεί σε αυτή την, ε, την παιδεία υπάρχουν, σε αυτούς, σε αυτούς τον τομέα. Και αυτό είναι η εφετηρία, το είπατε και εσείς η ίδια. Σήμερα έχουμε κάποια πράγματα τα είναι πετυχημένα όσον αφορά την διεθνή συνεργασία στην ανώτατη παιδεία. Έχουμε και σε άλλους τομείς όμως ε, τέτοια προγράμματα. Άρα θα πρέπει να το δούμε έτσι. Τώρα όσον αφορά την πρόταση του να ισχύει και εδώ ότι κάνουμε σε διεθνέ επίπεδο στην Ευρωπαϊκή, το κάνουμε και στην επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το πρώτο είναι ότι τώρα σε αυτή την πρόταση που εδώ συζητούμε, αλλά και στην πρόταση για τα μέσα τέτοια χρηματοδότηση, δεν θα ζητηθούν πολλά χρήματα. Εάν θέλετε κάτι να κάνετε, τότε θα πρέπει να πάρετε τα χρήματα από τα να βρείτε από αλλού κάποια χρήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε και προκειμένου η αύξηση που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την διεθνή επιτυχία δεν είναι το κάτι το τόσο φιλόδοξο όσο η πρόταση για το πρόγραμμα Έρασμος που είχαμε ζητήσει 70% ενώ για την εξωτερική διάθεση μόνο 10%. Και αυτό γιατί σπανίζουν οι πόροι, πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη τώρα. Όσον αφορά την πραγματικότητα για τον κλάδο, σαν τα παιδεία υπάρχει παράδοση συνεργασία. Σαν τα παιδεία έχουμε εκδρήματα τα οποία είναι τα ίδια περίπου παντού να ισχύει το ίδιο σε άλλους τομείς. Άρα θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και γι' αυτό είπαμε ότι και το Συμβούλιο πρότεινε τέτοιου συνεργασία. Όχι τόσο κινητικότητα όσο συνεργασία. Σε σχέση με τις νέες χώρες, το ίδιο Έτσι θα καλυφθούν και οι καινούργιε χώρε. και άρα όσο αφορά το PGA έχουμε αυτές τις τρίτε χώρε οι οποίε θα μπορούσαν να συμμετάσχουν αλλά δεν εδώ συμμετάσχουν ανέξοδα όπω είπατε γιατί θα πρέπει να αναπτύξουν δυνατότητες διαχείριση αυτών των πόρων. Και όπως είπατε και εσείς, υπάρχει το ζήτημα του τιμήματος που κανείς πληρώνει για την πολιτική απόφαση να συμμετάσχει. Όμως θα πρέπει αυτό να γίνει όσο ξεκάθαρο γίνεται, όπως το είπατε και στην, ε, στο εγγραφό σας, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, το πιο ωραίο τμήμα, τα εφαρμοστικά μέτρα και τις κατεξιδότητες πράξεις. Εδώ ισχύει ο πρώτος κανονισμός. Μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε και ισχύει στο νέο δημοσιονομικό οργανισμό είναι ότι τα ετήσια προγράμματα θα αποφασίζονται μέσω ε, μέτρων τέτοιων. Όμως, όταν λέμε εδώ για σκοπούς, δεν μιλάμε για τους συγκεκριμένους σκοπούς του προγράμματος. Θα πρέπει να δοθεί ορισμός μέσω των κατεξοδότηση πράξεων ή μέσω των ορισμών, ενώ τους συγκεκριμένους σκοπούς του, προγράμματος. Οπότε πολιτικής το περί των λεπτομεριών, των λειτουργικών στόχων, επιχειρησιακών στόχων του προγράμματος. Βεβαίω και υπάρχουν στόχοι πολιτικής και αποφασίζουν οι πολιτικοί. Όμως όταν είχε τη ώρα αυτό να μετατραπεί σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους, αυτό θα γίνει μέσω του προγράμματος μέσω της επιτροπολογίας πιστεύω. Δεν προχωρώ. Στα αυτά που συζητούμε για την επιτροπή του προγράμματος πιστεύω ότι και αυτό θα γίνει βάση των ρητρών επιτροπολογίας για τη φορολογία θα πρέπει να μην λύσουμε εδώ όλα αλλά θα πρέπει να ξέρω ότι θα δοθούν κάποιες υποτροφίες και για την ιδιωτική χρηματοδότηση ο τρόπος που παρουσιάζεται τα πράγματα είναι πολύ ρεαλιστικός. Και όσον αφορά τι εθνικέ αρχέ, τι εθνικέ υπηρεσίε, νομίζω αυτό το είπαμε την τελευταία φορά. Έχω μόνο μία παρατήρηση. Το είπα την τελευταία φορά, το ξαναπώ. Ανεξαρτήτω τη τελική λύση, ανεξαρτήτω του κατά πόσο νομιμότητα ή όχι, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σαν ελάχιστο είναι να εξασφαλίσουμε ότι ακόμη και αν δεν έχουμε ενιαίο συντονίζοντο φορέα ή μηχανισμό να έχουμε τουλάχιστον ένα τέτοιο διαγωνισμό τόσο ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον σε κράτο μέλο η, η εφαρμογή είναι, είναι... Αυτά όσον αφορά το προβλημα τώρα. Είπαμε σαν ελάχιστο να εξασφαλίσουμε κάποιο είδους αυθόρμητη επιτόπου μέθοδο συντονισμού Αλλιώς, αντί για απλούστευση θα έχουμε περισσότερες περιπλοκές. Αν χρειαστεί, να πάμε σαν το λόγο και σας τα ξαναλέω τα Ευχαριστώ κύριε Κορέλ. Το Σεπτέμβρη θα συζητήσουμε εντατικά για το ορατό και αναγνώσιμο και το καλά ορατό πρόγραμμα. Όπως ξέρετε όλοι το σχέδιο έκθεσής μου θα το υποβάλω το Σεπτέμβρη και όλοι θα έχετε την δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες εφόσον θα χρειάζονται ακόμα και τότε, τότε για να ψηφίσουμε το Νοέμβριο. Δεν νομίζω ότι θα δώσουμε το λόγο στην ε, Προεδρία γιατί θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Υπουργό σας για να μην ε, κάνουμε διπλή δουλειά. Θα ε, ζητώ την κατανόησή σας εδώ. Κλείνω τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Τα δύο έγγραφα, το σημερινό και το εκείνο της περασμένης φοράς, μην το βάλετε στα χρονοτούλαπα, ε, δείτε το για να κάνετε και τη σκέψη σας πάνω στο θέμα. Να προσθέσω κάτι. Ήθελα την άδειά σας να έχουμε αύριο το απόγευμα, ελεύθερο ίσως, θα δουλέψουμε ταχύτερα και δεν θα συνεδριάσουμε αύριο το απόγευμα. Ήταν έτοιμα που εξέφρασαν κάποιοι από εσά και κοίταξα να τα καταφέρω. Ελπίζω να συμφωνήσετε όλοι. Ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που είναι το πρόγραμμα για τη δημιουργική Ευρώπη. Creative Europe Program. Ζητώ συγγνώμη την Κομισιόν, ε, δεν έχουμε χώρο για όλους εδώ. Πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές τώρα για τη δημιουργική ναι, να περιμένουμε να να αλλάξουν τις θέσεις όσοι πρέπει. So. Everybody, especially the visitors, please take a seat or go out. Λοιπόν, παρακαλώ να καθίσετε όλοι, ειδικά οι επισκέπτες, με ησυχία, ή να εγκαταλείψουν την αίθουσα ή να καθίσουν. Wir haben heute das Programm... Äh, Σήμερα λοιπόν έχουμε κανονικά στην ημερήσια διάταξη για πρώτη φορά το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και η κυρία Κώστα είναι η συγγήτρια. Έχουμε κάνει ακρόαση που είχε μεγάλη απήχηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να αναφέρω τρία σημεία από αυτή την ακρόαση. Η διάφορα, τα διάφορα χαρακτηριστικά ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τα μέσα κλπ. Είναι σημαντικό να μην χάσουμε ε, επωνυμίες ε, καταξιωμένες, ιδιαίτερα το πρόγραμμα Media για τα ΜΜΕ. Τρίτον, το πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη σημασία των, ε, του μη κέρδους να μην επικεντρώνεται μόνο στα εμπορικά προγράμματα του κλάδου. Αυτά ήταν τρία σημεία που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της τελευταίας εκδήλωσης. Η κυρία Κώστα λοιπόν θα μας παρουσιάσει για πρώτη φορά τις εντυπώσεις της, γιατί τα προγράμματα έχουν παρόμοια προβλήματα ε, με τις εκτελεστικές πράξεις, τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Κυρία Ντεκώστα, Σίλβια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, πιστεύω ότι αυτή, αυτό το πρόγραμμα της Δημοτικής Ευρώπης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όντως εντάσσεται ε, σε ένα πολύ μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπως κατεδείχθη άλλωστε και από την ακρόαση που οργανώσαμε αλλά και από επαφές που είχα σε διάφορα επίπεδα. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ε, κατανοεί ότι και, καταγράφει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια προσπάθεια για καινοτόμα πρόταση η οποία δεν θα αφορά μονάχα τα μέσα επικοινωνίας και τον πολιτισμό αλλά και άλλα στοιχεία. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τους συναδέλφους με τους οποίους ήρθα σε επαφή σε αυτήν την πρώτη άτυπη συνάντηση που είχα και με τους ε, σκιώδεις εισηγητές εισηγητέ και βεβαίω να ευχαριστήσω και την Γραμματεία της Επιτροπής. Ε, θα πω δύο πράγματα εξ αρχή. Πρώτον, δεν πρέπει να λησμονούμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι μαζί με το πρόγραμμα Έρασμος για όλους, με όποιο όνομα και θα έχει και μαζί ε, και με τον ορίζοντα 2020 ε, θα αποτελέσουν ένα, μια τριάδα προγραμμάτων ε, που θα αυξήσουν κατά κάποιο τρόπο τον προϋπολογισμό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και τα τρία μαζί βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα μήνυμα αρκετά θετικό το οποίο ότι και το Συμβούλιο των Υπουργών ε, δεν θα αρνηθεί, ε, διότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να είμαστε και πιο ε, συνεκτικοί και με όλες τις πολιτικές οι οποίες αφορούν και την έρευνα και την καινοτομία και τον πολιτισμό, έτσι ώστε να έχουμε αυτήν την επιδιωκόμενη ανάπτυξη της γνώσης και την βιώσιμη ανάπτυξη της γνώσης μαζί με την κοινωνική ολοκλήρωση. Ε, είναι σημαντικό που εδώ ε, ε, γίνεται πιο τυπική η ενσωμάτωση ε, του ε, πολιτισμού καθώς επίσης ε, και, των, και της δημιουργικής πολιτιστικής βιομηχανίας με πιο επίσημο λοιπόν λέω τρόπο έτσι ώστε να φτάσουμε στους 12 τομείς παρέμβασης από performing arts μέχρι μουσεία, μέχρι αρχιτεκτονική κτλ. Δηλαδή μία σειρά ε, τομέων που ε, οργανικά πλέον εντάσσονται στο σύνολο του προγράμματος. Τρίτη σκέψη που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Βρισκόμαστε σε μία φάση όπου έχουμε αφενός την πρόκληση του διαδικτύου, την ψηφιακή δηλαδή ε, πρόκληση, ε, μέσα στην οποία εντάσσονται διαφορετικοί τρόποι παραγωγής, διαφορετικοί τρόποι διανομής ε, στις αίθουσες κτλ. Και ένα άλλο σκέλος το οποίο αφορά την εφαρμογή της ψηφιοποίησης ε, στην ε, πολιτιστική κληρονομιά, τη διατήρησή της ε, και την καινοτόμα αντιμετώπιση της. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και από το δημόσιο και από το ιδιωτικό τομέα μεγαλύτερη παρέμβαση έτσι ώστε έστω και μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης ε, να έχουμε αύξηση ε, της χρήσης, της κατανάλωσης, ας πω, εντός εισαγωγικών βεβαίως η λέξη κατανάλωση. Ε, καταλαβαίνουμε και διαπιστώνουμε ότι, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πολιτιστικά αγαθά σε όλους τους τομείς. Επομένως, ε, λέγεται ότι ο τομέας αυτός είναι αντικυκλικός από οικονομική άποψη ε, και που βεβαίως είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί ε, να δημιουργήσει καλύτερη ανάπτυξη και βεβαίως να έχει και αντικτύπω στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή ο τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Ε, και ε, έχουμε και τον τομέα της μεταποίησης ε, που οδηγεί σε νέες πρωτόγνωρες προκλήσεις ε, ε, και βεβαίως υπάρχει και αυτό το πολύ περίπλοκο ζήτημα το οποίο εγώ δεν θα ήθελα να θίξω που αφορά την προστασία των πνευματικών διανοητικών δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση ε, θεμάτων όπως είναι ας πούμε η πρόσβαση του Εβραίου κοινού στα πολιτιστικά αγαθά ε, την ε, ε, τον οικονομικό αντίκτυπο της πρόταση αυτής κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι τους τελευταίους μήνες και μετά την πρόταση της Επιτροπής σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μικρότερων επενδύσεων το δημόσιο τομέα και μικρότερων επενδύσεων μέσω των διαφημίσεων. Αναφέρομαι κυρίως ας πούμε στην τηλεόραση, αλλά ισχύει και για το κινηματογράφο. Αυτό σημαίνει βεβαίω, ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να σκεφτεί ότι αυτή η χρηματοδότηση είναι ικανοποιητική, αλλά 1,8 ε, δις για τον τομέα αυτό πιστεύω ότι είναι το απολύτως απαραίτητο και βεβαίως ε, καλό θα ήταν να μπορέσει να αυξηθεί και βεβαίως καθόλου να μην μειωθεί. Μία τελευταία σκέψη. Αναφέρεται στο κείμενο ε, της ε, Δημιουργικής Ευρώπης, αλλά με ασθενή τρόπο κατά την άποψή μου. Αναφέρεται λοιπόν ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να σεβαστεί και τις νομικές ε, βάσεις ε, της συνθήκης της Αμβονός και της ε, συνθήκης ε, της UNESCO και βεβαίως θα πρέπει να μπορέσει να ενσωματωθεί και στα άλλα υφιστάμενα προγράμματα. Κατά την άποψή μου αυτά τα σημεία θα πρέπει περαιτέρω να ενδυναμωθούν γιατί δεν αναφέρονται αρκετά σε ικανοποιητικό βαθμό. Όλο το πρόγραμμα προσανατολίζεται κυρίως προς ένα στόχο και προς ε, ε, μια γλώσσα αν θέλετε πιο οικονομική και βιομηχανική η οποία όμως δεν μπορεί ε, να καλύψει τον συνολικό ορίζοντα του πολιτισμού ας πούμε δεν υπογραμμίζεται και αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση που κάνω σαν εισηγήτρια και αυτό άλλωστε κατεδείχθηκε από τις ακροάσεις μας δεν καταδεικνύονται λοιπόν δύο μάλλον σημαντικά στοιχεία ε, της νομικής βάσης που βρίσκονται στις συνθήκη της Λισαβόνας, ε, ε, κυρίως η οριζόντια διάσταση του πολιτισμού, ο εγγενής χαρακτήρας και η εγγενής αξία του πολιτισμού στην Ευρώπη βάσει της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας αλλά και βεβαίως της άειλης και μη άειλης πολιτιστικής κοινωνίας Ευρώπης δεν αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία αυτά. Κατανοώ βεβαίω ότι γίνεται λόγο και αυτό είναι θετικό, αλλά ε, δεν μπορεί να βλέπουμε τα στοιχεία αυτά μόνο με όρου οικονομική ανταγωνιστικότητα. Και το άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να θίξω και είναι πολύ σημαντικό είναι η ενσωμάτωση ε, με άλλα υφιστάμενα προγράμματα. Κατά την άποψή μου δεν αρκεί να ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια καλή συνεργασία και καλή συμβατότητα με προγράμματα όπω το ε, Horizon 2020 κτλ θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες ε, αρχές ε, οι οποίες με αυτό τρόπο θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν ε, αυτά τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα τα οποία δεν καλύπτουν όμως το εύρος της πρόκλησης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αναφερθούμε μονάχα ε, σε αυτούς ε, τους πόρους ε, και σε αυτά τα εργαλεία. Στον ορίζοντα 2020 και στον, στην ευρωζωνική μάλλον ψηφιακή ατζέντα δεν εμφανίζεται σαφώς η έννοια του πολιτισμού όπως παλιότερα. Βεβαίως δεν είναι το αντικείμενο αυτό της εκθεσής μου, αλλά παρόλα αυτά ε, και μέσα από τροπολογίες ε, από άλλες επιτροπές βλέπω ότι θα πρέπει ε, να γίνει αναφορά σε αυτήν την εγκάρσια αντιμετώπιση του πολιτισμού. Το λέει και πριν η Πρόεδρος και στην ακρόαση κατέστησα φες ότι υπάρχουν κοινέ προκλήσεις, κοινά διακυβεύματα ε, και είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια επιλογή αρκετά δραστική ε, στα merging programs, ε, δηλαδή συγχώνευση προηγουμένων προγραμμάτων που αφορούσαν την επικοινωνία και τον ε, πολιτισμό σε ένα ενιαίο και μοναδικό πρόγραμμα. Το ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θίξω εδώ εγώ είναι ότι και οι αλυσίδε αξιών και τα business models είναι διαφορετικά στον πολιτισμό και τον δημιουργικό τομέα αφενός και τα μέσα επικοινωνία αφετέρου. Ενδεχομένως μπορούμε να προβλέψουμε κάποιες ενισχυμένες μορφές ε, αλληλεπίδρασης ε, και ε, αλληλοσυνεργασίας. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει στην διάρθρωση του προγράμματος να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό πλαίσιο νομικό, γιατί στο εσωτερικό του ε, υπάρχουν δύο διαφορετικά προγράμματα με διαφορετικό ε, τύπο διακυβέρνησης, με διαφορετικό προϋπολογισμό. Όπου από την μία ε, έχουμε τον πολιτισμό και την δημιουργική βιομηχανία και από την άλλη πλευρά τα μέσα ενημέρωσης. και επομένως το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο θα αφορά και, το, ε, και τους δύο τομείς, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος έτσι ώστε ε, οριζόντιες δράσεις να μπορούν να στηριχτούν. Επίσης πρέπει να πω ότι έλαβε υπόψη πολλές από τις προτάσεις, πολλά από τα μελήματα ε, τα οποία ε, ανέφερε και η ίδια η πρόεδρος ΠΑΚ όσον αφορά ε, και την απώλεια γνωστών επωνυμιών. Εμείς θα πρέπει να στηρίξουμε τις καταξιωμένες γνωστές επωνυμίες με συνειδητό τρόπο γιατί διαφορετικά ε, και οι εμπλεκόμενοι και οι ενδιαφερόμενοι θα χάσουν. Και η ίδια η διάρθρωση των δύο στοιχείων που συνυπάρχουν στο ίδιο πρόγραμμα ε, θα πρέπει να είναι ε, καθαρή. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί ο κάθε τομέας να παραμείνει αυτόνομος στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Και κάτι άλλο ήθελα να πω θα κάνω μία πρόταση προσανατολιστική κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι θέμα αρχή, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλω να ε, υποτιμήσουμε πολύ το θέμα και υποβάλλω το ζήτημα λοιπόν στην πρόταση, στην ε, ε, στην προσοχή σα. Δημιουργική Ευρώπη είναι ένα ωραίο σλόγγαν, είναι ένα ωραίο τίτλο που καλύπτει πολλά πράγματα όμως ε, με απασχολεί ε, το γεγονός της εγκατάλειψης της έκφρασης ε, πολιτισμού. Δεν, δεν γίνεται λόγο στην κουλτούρα, δεν γίνεται λόγο στον πολιτισμό και αυτό με απασχολεί λίγο. θα ήθελα λοιπόν να το υπογραμμίσω και να, να το βάλω έτσι λίγο στο κέντρο της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Όσον αφορά τώρα το θέμα της απόλυτης έλλειψης ε, στο κείμενο που ε, με ε, κατέπληξε. Δηλαδή η τοπική περιφερειακή διάσταση των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων που έχουν ε, στόχο ε, την ε, καινοτομία, την τοπική ανάπτυξη, διαπεριφερειακά προγράμματα που είναι πολύ σημαντικά και επίσης το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιφέρειες και περιοχές και πόλεις της Ευρώπης ο πολιτισμός ε, μπόρεσε να ε, δώσει εναλλακτικέ λύσεις σε περιοχές ε, όπου είχαν πληγεί από την αποβιομηχάνηση. Ας πούμε στη Λεκάνη του Ρούρ, στο Τωρίνο και σε άλλες περιοχές ο πολιτισμός έδωσε μία όθηση η πολιτιστική ανάπτυξη ε, μπόρεσε να ε, δώσει μια νέα επικέντρωση και μια νέα δύναμη ε, στις περιφέρειες και επομένως οι τοπικές αρχές μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές μπορούν να παίξουν πολύ καινοτόμο ρόλο. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό, νομίζω, και που νομίζω μάλλον ότι δεν ε, συνδέεται αρκετά, είναι το εξής. Ε, η λεγόμενη οικοδόμηση του ε, κοινού Υπάρχουν βεβαίως κάποια ποσοτικά στοιχεία στην πρόταση αυτή, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη αναφορά ε, στην κοινωνική διάσταση, ε, αυτή τη διάσταση των νέων κοινών ε, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, ε, οι ε, πολιτιστικές μειοψηφίες, ε, οι περιθωριοποιημένοι, γιατί βεβαίως εδώ μιλάμε όχι μονάχα για διεύρυνση ποσοτική, αλλά και εμβάθυνση ποιοτική του κοινού. Οι αναφορές οι οποίες βρίσκονται στον διατομιακό, στο διατομιακό τμήμα και που αφορούν την digital literacy ε, και την υψηλή κατάρτιση, οφείλω να πω ότι είναι πολύ γενικευτικές αναφορές και σίγουρα όχι ικανοποιητικές. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε τρόπους ε, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τις νέες γλώσσες, τους νέους τρόπους έκφρασης, να ενσωματώσουμε νέες ε, νέες, ε, νέα προγράμματα επαγγελματικά ε, έτσι ώστε να βρεθούν νέες καταρτήσεις αλλά και νέες δυνατότητες. Ένα άλλο σημείο το οποίο επανειλημμένα και σε άλλες περιπτώσεις το έχω αναφέρει είναι ε, η ε, ευρύτερη αναφορά στο θέμα της ε, κατάρτισης αλλά σε σχέση με τα πανεπιστήμια και σε σχέση με, τα, με τις καλές σχολές, τα προχωρημένα σχολεία κτλ. Και βεβαίως ο ρόλος των καλλιτεχνών και των δημιουργών δεν αναφέρονται σχεδόν ποτέ. Ε, αναφέρονται στα αγγλικά ως operators, αλλά αυτό, ξέρετε, μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η δημιουργική Ευρώπη ε, θα έχει έννοια μονάχα εάν υπάρχει συγκεκριμένο κεφάλαιο το οποίο θα αφορά ακριβώς τους δημιουργούς ε, και τους συγγραφείς και τους οι καλλιτέχνες ε, οι οποίοι ακριβώς είναι αυτοί οι οποίοι ε, θα στηρίξουν ε, αυτήν την πολιτιστική διάσταση. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να αποσαφινιστούν δύο πράγματα στους ορισμούς. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρώτον θα πρέπει να είμαστε ε, σίγουροι ότι θα αναφέρεται ο ορισμός του 2003, δηλαδή μικρές, μεσές, αλλά και ιδιαίτερα μικρές ε, επιχειρήσεις ή micro-enterprises, καθώς επίσης και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όχι τόσο για να υπάρξει ένα ειδικό κεφάλαιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτή τη στιγμή οι μικρές επιχειρήσεις του πολιτισμού, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, και οι φορείς φορείς ε, συνεργάζονται, αλλά θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης, ε, το operators ε, θα πρέπει να αποσαφινιστεί και θα πρέπει επομένως να πούμε ποιο θα είναι το προφίλ αυτών επί των οποίων γίνονται ή για τους οποίους γίνονται προτάσεις. Επίσης, ε, πολιτιστικά θεσμικά όργανα δεν αποσαφηνίζεται τι είναι αυτό ε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η νομική βάση δεν είναι ίδια, αλλά παρόλα αυτά ε, η πολιτιστική οργάνωση δεν είναι ούτε μη κυβερνητική οργάνωση, ούτε και απολύτως ε, ιδιωτική ας πούμε, επιχείρηση. Επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι ιδιαιτερότητες, ε, γιατί εδώ αναφερόμαστε σε δημιουργικότητα, σε νέους καλλιτέχνες κτλ. Να μην μπερδευτούμε. Υπάρχει άλλο ένα θέμα και εδώ μου θυμίζει λίγο και την κατάσταση με το Εράσμους Μόντους και τα λοιπά. Ε, προβλέπεται άνοιγμα μεγαλύτερο και αυτό είναι πολύ θετικό σε σχέσεις και διμερείς ε, με τρίτες χώρες, πράγμα που είναι πολύ θετικό και μάλιστα θα το επιθυμούσαν και οι ίδιοι οι operators. Άνοιγμα προς προς ε, επαφές και με μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις που δεν θα αφορά μονάχα την επικοινωνία αλλά και τις, ε, τα πολιτιστικά, τους πολιτιστικούς θεσμούς. Είναι, υπάρχουν χώρες μεμονωμένες οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή έχουν ε, ξεκινήσει δύσκολες εργόδεις ε, συνεργασίες, εταιρικέ σχέσεις με τη Βραζιλία ή με άλλες χώρες, αλλά στα πλαίσια αυτά υπάρχει δυσκολία όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Επομένως λοιπόν ορθότατα έχει προβλεφθεί αυτή η διάσταση του ανοίγματος προς άλλες χώρες 31 και μετά 37, τέλος πάντων είναι διάφορες ομάδες ε, χωρών. Όμως εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ε, δράσεις οι οποίες θα είναι ανοιχτέ σε αυτήν την διάσταση και αν θα ε, βασίζονται πάντα σε διμερείς επαφές ή εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίζει ανάλογα την περίπτωση πώς θα γίνονται οι συνεργασίες. Αυτό θα πρέπει να οριστεί καλύτερα. Ε, δεν έχει προβλεφθεί κανένα αποθεματικό του προϋπολογισμού ή κάποια επιπλέον γραμμή, γιατί απλώς γίνεται αναφορά στο άνοιγμα προς τρίτες χώρες. Ε, δεν θα ήθελα να είναι λευκή επιταγή. Όσον αφορά μάλλον κάτι άλλο, το γενικό κείμενο θέλει βεβαίως ε, να έχει έναν εγκάρσιο χαρακτήρα, αλλά συχνά ε, ε, παραμένει υπερβολικά γενικευτικό, υπερβολικά ασαφές τουλάχιστον σαν κείμενο κανονισμού ε, που δεν αποσαφηνίζει τις διαφορετικές παραμέτρους και όλες οι παράμετροι είναι ποσοτικές. Αλλά βεβαίως ε, ε, ο πολιτισμός και η δημιουργία πολλές φορές ε, αναφέρεται σε άειλα στοιχεία και επομένως δεν μπορούμε να αναφερθούμε μονάχα σε ποσοτικά στοιχεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει στα πλαίσια αυτά και με βάση και το δικό σας προτάσεων θα πρέπει να υποβάλουμε, λέω, και κάποιες αποσαφηνήσεις όσον αφορά το σημείο αυτό. Όσον αφορά τώρα τον προϋπολογισμό. Για τον προϋπολογισμό έχουμε πραγματικά αύξηση του 37% ε, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα. Έστω και αν βεβαίω ε, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ έχουμε περισσότερους τομείς και περισσότερες χώρες. Άρα τα ποσοστά δεν είναι τόσο ε, μεγαλύτερα. Πάντως στον κανονισμό αλλά μονάχα στο επεξηγητικό υπόμνημα ε, αναφέρεται η κατανομή του ε, προϋπολογισμού. Ε, όμως εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η κατανομή θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο σώμα του, κανονισμού με κλίδες κατανομής κτλ. και βεβαίως φαντάζομαι ότι μπορεί κάποια ευελιξία να υπάρχει στην ε, κατανομή αυτή, αλλά τουλάχιστον ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να καταγραφούν ελάχιστα ε, κατανεμόμενα ποσά. Όσον αφορά το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. γνωρίζουμε ότι είναι οριζόντιο για πολλά προγράμματα, επομένως δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Και εδώ γίνεται λόγος για ένα ευρωπαϊκό ταμείο ε, εγγυήσεων βάσει των οποίων θα γίνουν οι εθνικές ε, κατανομές. Θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα πορτφόλιο δανείων που από ό,τι λέγεται εδώ θα είναι ισορροπημένα στους διαφόρους τομείς αλλά δεν το ξέρουμε. Ε, εγώ συμφωνώ εάν αυτό δεν αντικαταστήσει αλλά απλώς προστεθεί στα κλασικά προγράμματα χρηματοδότησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφασιστεί να αποσαφινιστεί ε, και η γεωγραφική κατανομή. Οι νομικές βάσεις είναι διαφορετικές όσον αφορά ε, τα ε, δάνεια, το ξέρουμε αυτό, άρα θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε λίγο, να λίγο την κατάσταση. Είδαμε μονάχα δύο χρηματοπιστικά ιδρύματα τα οποία ήδη έχουν αντιδράσει θετικά, επομένως πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Το θέμα της ε, επιλεξιμότητας λοιπόν των δανείων θα πρέπει να αποσαφινιστεί περαιτέρω. Το γεγονός ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και του κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ο ίδιος ο κανονισμός δίνει κάποιους, ε, κάποιες κάποιους προσανατολισμούς ε, όσον αφορά το πορτφόλιο. Για τα desk, επαναλαμβάνω αυτό που ε, αναφέρθηκε και για το έρασμος, δηλαδή ότι υπάρχει το θέμα της, επικουρικού, της επικουρικότητας. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή, χωρίς αμφιβολία, ε, ο πιο σωστός προσανατολισμός δεν θα ήταν να δεχτούμε την advisor procedure που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς όμως να μπορούμε δηλαδή να μπούμε σε, ε, σε, σε λεπτομέρειες για τα ετήσια προγράμματα, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε ότι θα υπάρχουν κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, βάσει των οποίων θα μπορούμε να δούμε ε, και να υποδείξουμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Θα έχω κι άλλα να πω, αλλά τώρα δεν μπορώ, μου παίρνετε το λόγο. Ήθελα να δώσω κάποιες γενικές, ε, έτσι, να κάνω κάποιες γενικές προτάσεις, να δείξω κάποιους γενικούς ε, προσανατολισμού. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρο. Ε, Τρεις ζητούν το λόγο. Μπράγκο Καβαντά Σάκε. Κλείνουμε μετά. Θα μιλήσει η Κομισιόν. Πέντε παρατέταρτο το αργότερο πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα της αμνηστίας και να ακούσουμε και τον κύριο Κάβαντα. Και το, ε, όχι, τον κύριο Κα, ε, Τάκουλα μετά. Ε, κύριε Μπάγκο, σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μία ενημέρωση θέλω να κάνω. Ποτέ δεν ήταν απόλυτα σαφές αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Α, δεν κατάλαβα, δεν ε, μου είναι σαφές πώς θα γίνεται η διεύθυνση του προγράμματος για τις ΜΜΕ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα γίνεται η διαχείρισή του. Γι' αυτό εγώ απίφθηνα ε, ερώτημα προς την Κομισιόν και μου απάντησε λέγοντας ότι τα κονδύλια αυτά θα διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Επενδύσεων Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Καβαντά. Εισηγήτρια, συνάδελφοι, ευχαριστώ για όσα είπε σε Σίλβια και επίσης ευχαριστώ για όλα αυτά τα σημεία τα οποία έθιξες αλλά και τη συζήτηση που ήταν ενδιαφέρουσα. Αλλά και κάτι σε αρκετά και για μας είναι σημαντικό να ανταλλάξουμε τις απόψεις τόσο ώστε κάπως να οθήσουμε τα πράγματα όπως είναι σωστή κατεύθυνση και όπως είπατε κυρία Πρόεδρε Είπατε ότι έχουμε τρει ερωτήσει και γι' αυτό και νομίζω ότι είναι σημαντικό να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με το κείμενο το οποίο εδώ έχουν προ συζήτηση, διότι σε αυτά τα οποία είπα στις 6 Τετάρτου είπα ότι πήγαν τα πράγματα κάπως θολά ε, όσον αφορά το τι μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαμε διάφορα τα οποία έπρεπε να, α, έπρεπε να, να, να, να ε, διευκρινιστούν κύριε Πρόεδρε να σας πω κάποια πράγματα που έχω σε διαφορετική προτεραιότητα από εσάς όσον αφορά τα βασικά σημεία, να είμαι σύντομος, συνθετικός, ε, να σας πω τα εξή. πρωτα Πρώτα-πρώτα έχω ακόμα κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τον ορισμό του προγράμματος και σε σχέση με την πρικοδότηση που αφορά το καθένα από αυτά τα σύνορα που είπατε και όσον αφορά την συνάρθρωση αυτή ε, σε σχέση με τις διαφορετικές πτυχές του προγράμματος αλλά και τους πόρους που θα δοθούν. Ε, θέλαμε να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια, δεν την βρήκαμε. Τώρα όσον αφορά ε, αυτού του είδου το Ταμείο Εγγυήσεων που προτείνει η Κομισιόν, δεν μας τα είπε τόσο ξεκάθαρα, γιατί θα πρέπει από πλευρά ε, χρημάτων, θα πρέπει να μην έχουμε διασπάθησή τους και ε, σε όλους τους διαμέσους. Επίσης, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, δεν έχει κανενός είδου εγγύηση σε σχέση με την εκτέλεση θα πρέπει να αποσπάσουμε και τις εγγύσει, ιδίω μια από η σημερινή συγκυρία είναι συγκυρία κρίση και επίσης η δεύτερη φάση να σας πω και κάποια άλλα πράγματα που δεν θεωρώ ότι είναι και αμεληταία και να δούμε κατά πόσο μπορεί σήμερα ή κάποια στιγμή να μα διευκρινίσει η Κομισιόν όσον αφορά τον ορισμό των σκοπών του προγράμματος που είναι πάρα πολύ ε, ασαφής. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν καλύτερα και έτσι να ξέρουμε ακριβώς ο προπολογισμός τι θα καλύψει επίσης όσον αφορά την ε, συγχώνευση αυτών των γραφείων ε, ε, ενημέρωσης σε κάποιες χώρες, υπάρχουν προβλήματα μεγαλύτερα, υπάρχουν περιπλοκές. Πώς τα βλέπετε στα πράγματα, τι θα γίνει επίσης όσον αφορά την εποπτεία, όσον αφορά την εξολόγηση του προγράμματος, όλα αυτά κατά τη γνώμη μου επίσης επιδέχονται ξεκαθάρισμα. Τώρα να δούμε το ότι να... πέραν τον να δούμε τι διακυβεύεται από λόγες οικονομικής και να δούμε επίσης ποιοι θα είναι οι, όχι, όχι, οι πραγματικοί, οι τελικοί, οι λειτουργικοί ε, επιλέξιμοι, λειτουργικοί δικαιούχοι και όχι ενδιάμεση. Όχι, εγώ δεν θα δώσω λευκή δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και να εκτιμώ. Όσον αφορά αυτό το, τη Δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα, έχω την αίσθηση ότι τώρα βρήκαμε αυτή την ωραία έκφραση που είναι πάρα πολύ θετική, πάρα πολύ όμορφη αλλά εδώ τώρα καλύπτουμε κάτι πάρα πολύ θολό πλευρά τη Άρα που δεν μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φως και επίση όσο να κάτι άλλο το οποίο με ενδιαφέρει πολύ είναι το ότι το πρόγραμμα αυτό, η ε, Διεθνική Ευρώπη, καλύπτει δύο πραγματικότητε οι οποίε είναι πραγματικά τελείω διαφορετικέ και θα πρέπει να τι σεβαστούμε και τι δύο πρώτα-πρώτα το πρόγραμμα μέντια του, πόσο, πόσο, πόσο έχει πετύχει. Εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν επιδέχεται καμία κουβέντα. Γιατί όλα πάνε πάρα πολύ καλά, επομένω το αφήσουμε στην ησυχία του. Γιατί επομένω να πειράξουμε κάτι που είναι μια χαρά. Επίση, όσον αφορά το, τα, τα οπτικοακουστικά, το είπατε για παντού στην Ευρώπη, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πετύχει και όσον αφορά όλα αυτά, την, και τα πολιτιστικά και δεν καταλαβαίνω γιατί το πρέπει εδώ πέρα να περιπλέξουμε κάτι το οποίο λειτουργεί εδώ και τόσο καιρό και σας ξαναλέω γιατί θα πρέπει θα πρέπει να μπλέκουμε τα πράγματα γιατί έχουμε, έχουμε ξεκάθαρε ρυθμίσει στι δημοσιονομικέ και ξεκαθαρού στόχου. Ευχαριστώ. Τώρα επίση, όσον αφορά την εκτέλεση, νομίζω ότι θα, θα δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα, τι του βάθου να θα, θα γίνει. Σα ευχαριστώ καλά τα πήγατε και συνεχίστε εγωμένως τη συνεργασία πάντα με ανοιχτό πνεύμα, θετικά και έτσι να μπορούμε όλοι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε τελικά κάποιες, κάποια ξεκαθαρίσματα. Πρόεδρο. Η κυρία Σάκε, σύντομα και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ, ναι, είναι σύντομη και πιστεύω ότι πρώτα-πρώτα θέλω να σας πω πόσο θεωρείται είναι θετική αύξηση της ε, προοικοδότησης ε, λέμε πολλά για τον πολιτισμό όμως πάρα πολλέ φορέ. δεν έχουμε αυτή την αύξηση περιοδικότητας. Άρα τα πράγματα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και η κοινωνία των πολιτικών επίσης θα το δει πάρα πολύ θετικά και η πολιτική κύκλη, άρα θα πρέπει να πασχίσουμε να έχουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα, πολλές φορές να έχουμε αλλαγή της κουλτούρας ε, μέσα στους οργανισμούς και επομένως αυτή η μετακίνηση προς τα δάνεια είναι πάρα πολύ υγεία φαινόμενο, όμω θα πρέπει να επεξεργαστούμε τι λεπτομέρειε του χρηματοδοτικού μέσου. επίση ε, δεν μπορώ παρά να πω ότι είναι σωστά όλα αυτά που λέμε για λιγότερη αυτοκρατία, περισσότερη αποτελεσματικότητα και το να μιλούμε για μάρκε, ε, σήματα μάρκε τέλο πάντων. Ε, αυτό είναι ένα από τα πολλά. Ο κόσμο τη ουσία θα μα χειροκροτήσει τώρα να δούμε τι γίνεται με τι μικρότερε φορεί και να μην βλέπουμε μόνο τα εμπορικά βλέπουμε μόνο τα εμπορεύσιμα, προϊόντα, τα πολιτιστικά, αλλά να βλέπουμε και την αξία για όλο τον κόσμο, για τη δημόσια την αξία, την κοινή αξία. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει και με την ψηφιοποίηση και αυτό αξίζει να το εξηγήσουμε καλύτερα για να το δούμε στις λεπτομέρειές του. Χαιρετίζω επίσης ότι θεωρηθήκαμε ως παγκόσμιος παίκτη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις εξωτερικές δράσεις. Ίσως υπάρχουν προτάσεις. Ίσως και προτάσεις αυτές μπορεί να τις λάβει υπόψη η εισηγήτρια. Κινητικότητα, προσβασιμότητα, συνδυασμό διαφορετικών αποτελεσμάτων, επιπτώσεων, σκοπών που διώκουμε και πάντως κατακλείδη, να σας πω το ότι στα πλαίσια των εξωτερικών δράσεων θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ε, εκταμείευση το πόρο, πούμε, τα ταμεία της διεύρυνσης, για να καλύψουμε και ζητήματα πολιτισμού. Να, που μπορούν να ωφελήσουν οι πόροι που θα εκταμιευθούν για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο διευθυντής ε, του πολιτισμού έφυγε και πήγε σε άλλο τμήμα. Έτσι μου είπαν. Τώρα δραστηριοποιείται σε άλλο τομέα της ε, έρευνας. Δεν δίνω το λόγο στην διάδοχό του, αλλά στην υπεύθυνη. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όντως αποχωρεί ο διευθυντής και εγώ θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες διευκρινήσεις και κατόπιν η κυρία Σίλα θα σα πει τι γίνεται από πλευρά οπτικοακουστικών, αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τι παρατηρήσει. πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και τώρα έχουμε μια-δυο διευκρινησει πρωτα Πρώτα-πρώτα όσον αφορά το πόσο ε, διαφέρουν τα, τα θέματα στα πλαίσια του, στα πολιτιστικά. Γι' αυτό και το Δημιουργική Ευρώπη είναι ένα πρόγραμμα πλαίσιο, έτσι το ονομάζουμε. Και εδώ έχουμε διαφορετικές ε, ε, απολύξεις, διαφορετικές ε, επιπτώσεις ε, επιμέρους γιατί εδώ πέρα αυτές οι δέσμες, οι δέσμες αφορούν διαφορετικά μέσα, διαφορετικές, ε, ε, διαφορετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, άρα γι' αυτό θα πρέπει να στοχεύσουμε στους εμπλεκόμενους κατά παραγγελία κατά περίπτωση όσον αφορά τον τομέα των μη κερδοσκοπικών φορέων, πολύ σημαντικός, ιδίω όσον αφορά τα πολιτιστικά. Εγώ ασχολούμαι με αυτό και όπως βλέπετε ε, αυτό ήταν ο βασικό στόχο των μη κυβερνητικών φορέων. Με εξαίρεση κάποιε μεταφράσει. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να στοχεύσουμε στους εκδοτικούς οίκους και αυτοί μπορούν να ζητήσουν ε, κάποιο είδου ενισχύσεις και υποτροφίες μόνο στα πλαίσια των μη γεωδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Οι εταιρείε θα έχουν αλλού είδου διευκολύνσει όσον αφορά τι εκτελεστικέ, εφαρμοστικέ και κατεξοδότηση πράξει. Τα συζητήσαμε στα πλαίσια του Έρασμο για όλου και ο Τζορ Κορέλ σα είπε τι προβλέπει ο δημοσιονομικό κανονισμό. Παρ' όλα αυτά όλες οι βασικές πολιτικές πτυχές, όλες ορίζονται μέσω της νομικής βάσης, γενικοί στόχη και οι προτεραιότητες, κάτι το οποίο δεν είχε ισχύσει προηγουμένως στα πλαίσια ε, των πολιτιστικών κατά πολλού τρόπου, Περισσότερο από στο παρελθόν και κάποιους, κάποιους δείκτες που δεν υπήρχαν προηγουμένω. Τώρα, στον αφορά το ζήτημα τη εσωτερική αξία των πολιτιστικών. Συμφωνώ με τον είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όντω, αυτό δεν το έλεγε ρητός η πρότασή μας, εμεί θεωρούσαμε ότι, ότι υπονοείται. Οπότε, το πρόγραμμα αυτό θέλει να δημιουργήσει όσο γίνεται καλύτερο περιβάλλον για του ε, καλλιτέχνε, του φορεί του, διασυνοριακά να δρούν, να μπορούν να ελκύσουν, να αγγίξουν κόσμο παντού, ε, Βεβαίω και μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση και επίση νομίζω ότι ο πρώτο βασικό στόχο, η ποικιλομορφία, η πολιτιστική κλπ. είναι φυσικά πολιτιστικού χαρακτήρα. Δύο λόγια όσον αφορά την πολιτική, την περιφερειακή διάσταση αυτών των δραστηριοτήτων. Πρώτα-πρώτα επισύρω την προσοχή σα στο ότι μέσα σε λίγε εβδομάδε πρόκειται να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα πρόταση που θα αφορά τι ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτεύουσες για την περίοδο μετά το 2020. Πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που έχουμε αναπτύξει, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τοπικές, περιφερειακές, ευκαιρίε ανάπτυξη. Τώρα, όσον αφορά την δημιουργική Ευρώπη πιο συγκεκριμένα, επίση και τη δέσμη την πολιτιστική. Μιλάμε για Ευρωπαίο ε, πρόγραμμα, αλλά πρόκειται περί συνεργασία Ευρωπαϊκή, συμπληρώνουμε το τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Πάντω σα τονίζω ότι αυτή η νέα αιστεία τη προσοχή μα για το συγκεκριμένο κοινό αφορά του πολιτιστικού φορεί που προσπαθούν να εισδύσουν τοπικά για να είναι πιο αποτελεσματικοί τοπικά και οικονομικά και Εδώ πέρα το να βρούμε, το να δημιουργήσουμε στο στο κατάλληλο κοινό έχει σημασία και επίσης ε, σε σχέση με αυτό έχω να σα πω ότι σε σχέση πάλι με το πώς θα αγγίξουν περισσότερο κόσμο, νέους, ε, έτσι πρέπει να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, αυτό είναι ένα εργαλείο να καλύψουμε αυτούς τους παραμερισμένους, τους μη προνομιούχους, τους, τους περιθωριοποιημένους. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Πάροχη. Θα, θα πρέπει να δούμε τέλο πάντων στου ορισμού την ορολογία, να δούμε τι θα καλύψουμε από οργανισμού και από καλλιτέχνε. Τώρα για του ε, ορισμού, έχουμε την ε, σύσταση 2003 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ΜΜΕ, οπότε και έτσι θα καλύψουμε ένα σωρό ΜΜΕ αλλά και μικροεπιχειρήσει. Και εδώ μπορούμε να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά κάποιο μέτρησης, φακάλα λέτε μέτρηση, ο καλό λέτε ότι εδώ πέρα είναι καθαρά ποσοτικοί δείκτε ή τα κριτήρια. Αλλά εμεί θεωρούμε ότι αυτό το αξιολόγηση δεν είναι σημαντική η ποσοτική. Έχουμε τις αξιολογήσεις, σας παραπέμπω στο 14.3. Στο 14.3. Και σα διευκρινίζω ότι η μεθοδολογία σε όλα μας τα προγράμματα αφορούσε στο να θεσπιστούν για πρώτη φορά τέτοιοι δείκτες στην νομική βάση για τους ε, συγκεκριμένους αυτούς στόχους. Και όλα αυτά για να μπορούμε να δούμε τι συνέπειες υπάρχουν, να έχουμε, γιατί έχουμε αυτούς τους δείκτες τους ποιοτικούς επίσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε και να υπάρχει και ποιοτική αξιολόγηση. Τέλος, από πλευρά μου, Όσον αφορά την απόδοση ευθυνών για την δαπάνηση των πόρων, εδώ υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας, διαφάνειας, δημοσιότητος και επομένως λογοδοτούμε στην αρχή των προπολογισμών. Και τώρα δεν κοιτάει την έχει συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω απλώς ένα θέματα και για τα ΜΜΕ και κάτι άλλο για ε, το χρηματοδοτικό μέσο. Ένα από τα θέματα τα οποία ανέκυψαν είναι πάλι το ζήτημα των ορισμών και το ότι χρειάζεται να υπάρχει ακρίβεια, συγκεκριμένος χαρακτήρας των ορισμών και όταν λέμε πάροχος έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να καλύψει τους εν δυνάμει ε, επιλέξιμους φορείς εμπορικούς, δίκτυα κινηματογραφικά κλπ. Φεβείς και το χτενίσουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι καταξιωμένη συνταγή εις το παρελθόν. Δύο λόγια, ίσως λίγο παραπάνω, όσον αφορά τους, ε, την, την, το μέσο διευκόλυνση, το μέσο το εγγυητικό για για τους πολιτικούς φορείς που ξεκινάμε με την γεωγραφική κάλυψη και ένα από τα βασικά το οποίο πρέπει να σας αναφέρω είναι το εξή. Δεν δίνουμε τίποτα σε ομοτοπιστωτικά ιδρύματα. Απλώς είναι διτίθεται αυτό το ποσό για να καλυφθούν αυτοί έναντι του τι παρέχουν στου καλλιτεχνικούς φορεί. Και σε σχέση με το ότι ίσχυε στο παρελθόν, τώρα γίνεται χρήση πολύ λιγότερο από στο παρελθόν. Α πούμε το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και ε, Τέλο πάντων, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το χρηματοδοτικό μέσο σήμερα. Γιατί έτσι αλλάζουν οι νοοτροπίε. Και έχουμε κάνει βήματα πρόοδου τι τελευταίε εβδομάδε. Υπάρχει τα αποτελεσματική συμφωνία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Και Μπορούμε να σα δώσουμε περισσότερε λεπτομέρειε για το πώ λειτουργούν τα πράγματα. Και έτσι το σχετικό κομμάτι του, του κανονισμού να είναι σαφέστερο. Ξέρουμε επομένω ότι χρειάζεται την ΕΕ να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κρατικά στι τράπεζε. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Και βεβαίω θα δώσουμε το Κοινοβούλιο επιπλέον πληροφορίε, αλλά και στο Συμβούλιο. Και σα ευχαριστώ. Για τα ΜΜΕ όμως δεν είπατε τίποτε. Για τα ΜΜΕ τι θέλατε να πείτε, δεν τίποτε. Ευχαριστώ για τις διάφορες επιχειρήσεις, τους δραστηριοποιούμενους αν θέλετε στον τομέα. Α, και για την επωνυμία. Η επωνυμία του ΜΜΕ είναι γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Ταινίες κινηματογραφικές που διανέμονται με το λογότυπο του, των ΜΜΕ έναντι αυτών χωρίς το λογότυπο, βλέπουμε ότι οι πρώτοι ε, επιτυγχάνουν υψηλότερη τιμή αν πρόκειται να ε, χρηματοδοτηθούν. Οπότε επηρεάζει την αγορά η επωνυμία. Άρα λοιπόν, γιατί δεν το είπατε, θα το πω εγώ. Η επωνυμία θα διατηρηθεί. Το brand name θα παραμείνει. Ε? αν είναι επωνυμία όπως μας είπατε, θα παραμείνει και τα επόμενα έξι χρόνια έτσι θα είναι. Όχι, η προσέγγιση της Κομισιόν είναι ότι ε, αν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ε, από νομική, στη νομική βάση, το, ο νέος λογότυπος της Κομισιόν θα είναι επίσημη ταυτότητα για όλα τα προγράμματα, αλλά το όνομα θα παραμείνει για τη δέσμη. Είναι, είναι περίπλοκο. Είναι περίπλοκο. Μα είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή επανεφευρίσκεται τον τροχό. Αντί να κρατάτε αυτά που είναι καλά, λέτε το media program έχει εισαχθεί, το ξέρουν όλοι, το λογότυπο το ξέρουν. Και γι' αυτό ο κύριος Κάβαντα και εγώ δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί δεν μας έδινε απάντηση ο προηγούμενος. Τώρα μας δίνεται, αλλά καταλαβαίνουμε και τι θέλει η Κομισιόν. Το λογότυπο του Μίδια δεν μπορείτε τώρα να το αλλάξετε, να μην υπάρχει πια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι, κυρία Ντεσίλβα, τι να κάνουμε. Ε, με σας πρέπει να τα πούμε, αφού ο κύριος Σούρα έφυγε και τώρα θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε με εκείνους που έκαναν τη δουλειά και ίσως δεν θέλανε να την κάνουν και δεν συμφωνούσαν με αυτό που έγινε. Επανέρχομαι. Μπορείτε να διευκρινίσετε στην Κομισιόν ότι το η επωνυμία είναι επωνυμία και το media είναι κάτι που έχει ένα λογότυπο που φαίνεται σε κάθε ταινία και δεν θα φαίνεται στο μέλλον. Δηλαδή θα ξεχνάμε το, το παρελθόν και θα αφήνουμε να το λησμονούν και οι άλλοι. Ε, αυτό είναι πραγματικά άσχημο. Θα δώσουμε και στην κυρία Κώστα το, το λόγο για να... Αλλά προηγουμένως θα, ναι, θα απαντήσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πακ. Θα είμαι όσο πιο σαφής μπορώ και μετά εσείς θα συνάγετε τα συμπεράσματά σας. Η προσέγγιση της Κομισιόν είναι ότι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το λογότυπο του Media μέχρι το τέλος ε, των δημοσιονομικών αυτών προοπτικών. Από τις επόμενες δημοσιονομικές και μετά μόνο επωνυμίες που ε, εντοπίζονται και έχουν αναγνωριστεί ως ε, επωνυμίες στη νομική βάση του προγράμματος θα χρησιμοποιούνται. Έχουμε και το Media Strand, τη δέσμη Media που θα μπορεί να χρησιμοποιεί την οπτική ταυτότητα και η νέα οπτική ταυτότητα της Κομισιόν θα χρησιμοποιείται παντού, εκτός και αν αναφέρεται ρητός διαφορετικά, κάτι διαφορετικό στη νομική βάση. Ε, αυτό είναι. Να δούμε, θα δούμε τότε και εμείς μήπως μπορούμε να αλλάξουμε τη νομική βάση. Ναι, ναι, νομίζω διευκρίνηση γιατί την άλλη φορά εδώ είπαμε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο, οπότε δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και κυρία Σίλβα που είπε την αλήθεια. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι, ε, προβληματίστηκε και όπως προείπαμε, Θέλαμε ακριβώ να πάρουμε το διευκρινήσει, οπότε και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό πρόκειται να πείσει στου συναδέλφου. Οπότε νομίζω ότι Πρόκειται κατά αυτόν τον τρόπο να σημειώσουμε πρόοδο και θα πρέπει να εξεταστεί πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο προγράμματα σε σχέση με ε, αυτές τις δύο δέσμες. Και πάντως, συζητά αφού είπε ο κύριος Μπάγκο, Σας ε, διαβεβαιώ. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε. και το είπε και άλλωστε και Επιτροπή, το Κοινοβούλιο. Θέλουν, θέλει και εκείνο να εμβαθύνουμε. Πρόκειται για μια καινοτομία. Και νομίζω θα προκύψουν πολλά, θα διευκρινιστούν πολλά. όσον αφορά για την ισορροπή λύση που θα πρέπει να δώσουμε και να μην έχουμε μόνο τις μεγάλες αλλά και τις μικρές εταιρείες να καλύψουμε που να μπορούν όλοι αυτοί να έχουν λοιπόν πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης. Δεν θέλουμε να καταρχίσουμε ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως, θέλουμε να το συμπληρώσουμε. Γι' αυτό σας λέω. ΜΜΕ θα τα πάνε καλύτερα και έτσι θα έχουμε περισσότερε δραστηριότητε από πλευρά των ΜΜΕ, περισσότερε Δυνατότητε που θα του δοθούν. Έτσι θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Επομένω θα πρέπει να κάτσουμε να δώσουμε κάποιου καλύτερου ορισμού στον οργανισμό. Θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο. Κύριε Καβαντά, παρουσιάσατε το πώ έχουν τα πράγματα απλώ προδρατήτων. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτά τα οποία τονίσατε θα τα ξαναδούμε. Όλα αυτά τα οποία τονίσατε, όλα αυτά εγώ τα καλύπτω. Πάντω θα κάτσω να συνεργαστώ μαζί σα και να δω πώ θα τα κάνουμε καλύτερα. Τώρα, θα ήθελα και εγώ να σα πω ότι έτσι θα δώσουμε ένα μήνυμα, ένα θετικό μήνυμα. Όμως θα πρέπει για να αντιμετωπιστούμε στην, ευρωπαϊκή πρόκληση όλα αυτά τα οποία συζητούμε να τα βάλουμε σε όλες μας τις πολιτικές. Θέλουμε περισσότερη αγωνιστικότητα, θέλουμε περισσότερες δυνατότητες να αποκτήσουμε. Αυτή είναι η πρόκληση που γίνεται αυτό το πρόγραμμα και παραπέρα. Ξέρετε ότι τα πολιτιστικά έχουν δυτή φύση και πολιτιστική και οικονομική. Μάλιστα μέσα του πολιτισμού τονίζεται και η οικονομική ενταγνωστικότητα. Τα είπαμε. Ακούσατε και τις δικές μου προτάσεις. Επίση, όσον αφορά τον ορισμό των ΜΜΕ, να δούμε τι έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. εδώ πέρα μιλούμε για τι επιχειρήσει, θα πρέπει να καλύψουμε και τι μικροεπιχειρήσει. Τώρα, άλλο. Για τη διαφάνεια όσον αφορά την διάθεση των πόρων. Για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Μια που μέσω της ε, επικουρικότητας μπορούμε αυτά τα γραφεία να τα ενισχύσουμε. Να κάνουμε πρόσκληση υποβολής προσφορών γιατί θέλουμε τα κριτήρια να είναι σε όλες τις περιπτώσεις σαφέστερα να έχουμε μια κυκλική αναλλαγή των εμπειρογνωμόνων, είναι σημαντικό και το αποτέλεσμα αυτής της, υποβολή, της πρόσκλησης προσφορών θα πρέπει να γίνεται προς του ενδιαφερομένους. Προσοχή. Να είμαστε συνεπείς στις απαντήσεις στα ερωτήματα. Για όλες τις χώρες. Ελπίζω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία και στο μέλλον είδαμε βεβαίως ε, και την ε, ε, μερική συμφωνία του Συμβουλίου των Υπουργών. Εγώ είχα συνάντηση και με την ε, Δανέζικη Προεδρία αλλά και με τον επιτετραμένο πολιτισμό <coughs> της Κύπρου ε, και πραγματικά πιστεύω ότι η Κομισιόν θα την ευήκονους έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε μια καλή δουλειά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος και καλή συνέχεια σας εύχομαι. Μάλιστα. Πάμε στο σημείο 6 η Ευρώπη για τους πολίτες. Ε, Χάνου, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν νομίζω ότι θα μακρηγορήσουμε εδώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος με βάση κάποιες σημειώσεις μου. Το θέμα της νομικής βάσης είναι ανοιχτό ακόμα, να το συζητήσουμε και θα δούμε τι θα βγει στην πάλι αυτή με την Κομισιόν. Ελπίζω να είναι καλό το αποτέλεσμα και να κατησχύσει η λογική. Και παλιότερα ε, ως εισηγητής για το πρόγραμμα είχα δραστηριοποιηθεί, για το πρόγραμμα αυτό ως εισηγητής, το πρόγραμμα ήταν καλό, το feedback ήταν καλό και γι' αυτό ελπίζω ότι και η Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, το βλέπουν ως επιτυχημένο πρόγραμμα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τους βοηθούς που παρευρέθησαν. Είχαμε ενιαίες απόψεις για τα θέματα και είναι καλό να ακούσουμε και από την Πρόεδρο και από άλλους όμως τις απόψεις τους Επί ορισμένων θεμάτων λοιπόν θέλω να ακούσω τη γνώμη των άλλων και θυμίζω ότι συζητάμε το σχέδιο του Συμβουλίου. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και τις απόψεις της Κομισιόν και πώς συνδέονται με, το, του Συμβουλίου και σε ποιο βαθμό άλλαξαν κάποιες θέσεις. Πρώτον, ο, το, ο στόχος πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή κληρονομιά και ο βελτιωμένος αναβαθμισμένος ρόλος της. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο θέλουν να αναβαθμίσουν την ιστορική ε, συνείδηση. Ε, ένα πρόγραμμα όπως ένα σπίτι πρέπει να έχει καλά θεμέλια και το θεμέλιο σε αυτό το πρόγραμμα που θεωρείται στέρεο είναι ε, ε, η ιστορική μνήμη. Θα πρέπει λοιπόν από κάτω προς τα πάνω να οικοδομηθεί το πρόγραμμα με πρωτοβουλίες σημαντικές, νέες πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρουν και νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Και όταν θα προχωρήσουμε και θα αναπτύξουμε το θέμα αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει και διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού, ώστε νέα καινοτόμα προ... projects, έργα με σαφή ευρωπαϊκή προοπτική να συνδέονται και με τα παλιά προγράμματα. Θέλω εδώ να ακούσω και την γνώμη των συναδέλφων, πώς το βλέπουν και τι ποσοστό θα πρέπει να ε, δοθεί στις μικρές πρωτοβουλίες και στα μικρά προγράμματα και έργα. Ένα κεντρικό στόχος ήταν ότι δεν πρέπει να είναι πρόγραμμα ελίτ, ελιτίστικο πρόγραμμα. Πρέπει να είναι πρόγραμμα για τους πολίτες και ε, τελ, επίσης διαπιστώνεται στο τρίτο άρθρο ότι τα υπόροι για τα ΜΜΕ θα πρέπει να ε, καλύπτουν και γενικότερες ενημερωτικές δραστηριότητες που αφορούν και τους στόχους της Ένωσης. Βέβαια, ο προπολογισμό για αυτό το πρόγραμμα είναι σχετικά μικρός. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πεπισμένο ότι δεν πρέπει από αυτό το μικρό πρόγραμμα να διαθέσουμε μικρά κονδύλια στην Κομισιόν για άλλες επικοινωνιακές στρατηγικές. Αυτά τα μέσα, αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος και για ενημέρωση στα πλαίσια του προγράμματος το κόστος, ε, οι δαπάνες θα πρέπει να είναι ε, όσο γίνεται πιο χαμηλές. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη να έχουν μια ευρεία αυτονομία και στην εφαρμογή των ε, προγραμμάτων. Όλοι πιστεύουμε ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη, αμοιβαία και βεβαίως ο έλεγχος, ίσως ο έλεγχος γενικά είναι καλύτερο, να είναι καλύτερος από την εμπιστοσύνη, αλλά χρειάζεται και εμπιστοσύνη. Και αν ε, ελέγχονται υπερβολικά οι πρωτοβουλίες των πολιτών, ε, μπορεί να καταστραφεί το πνεύμα αυτών των πρωτοβουλειών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και στο, ε, στην τωρινή προγραμματική περίοδο Μάλιστα, ε, μικρές πρωτοβουλίες έγιναν ε, μεγάλες επιτυχίες, ακριβώς επειδή υπήρχε ε, στην προηγούμενη περίοδο εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω και απόψεις των συναδέλφων. το χρονοδιάγραμμα είναι ότι στις 15 Σεπτεμβρίου θα δοθεί συνέχεια στο θέμα αυτό. Μέχρι τότε θα συζητούμε και θα ετοιμάσουμε και τυχόν τροπολογίες και η Κομισιόν και το Συμβούλιο εν τη σοφία τους ελπίζω να υποστηρίξουν και να δεχτούν τις προτάσεις μας. Μάλιστα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, και όπως αποφασίσαμε, θα έχουμε διαδικασία συναπόφασης όπως μας συνεβούλευσε η νομική μας υπηρεσία. κύριος ε, Ρέπο ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μιλήσαμε και για το Εράσμους σήμερα και μάλιστα λυπάμαι που δεν πρόλαβα να έρθω. Ήμουν στην Ίμκο. Αλλά θα υποβάλω γραπτό ερωτήσεις στην Κομισιόν. Εγώ Είμαι σκιώδης ε, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και πιστεύω και εγώ ότι η νομική βάση έχει γίνει πια μια φάρσα. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για δραστηριότητες και για συμμετοχή ότι θα πρέπει να ακούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της ουσίας. Τρία σημεία θέλω να τονίσω. Την περασμένη εβδομάδα επίσης δεν ήμουν παρόν στη συνεδρίαση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ίσοι όροι συμμετοχής για όλους. Μιλώ εδώ για περιφερειακές περιοχές, απόμακρες και βέβαια θα πρέπει να δούμε και την ε, ίση κατανομή των πόρων. Θα ήθελα να εξετάσουμε τα πραγματικά κόστη εδώ, ούτως ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα προγράμματα σε όλες τις χώρες. Αν και νομίζω ότι δεν επαρκεί ένα πρόγραμμα ανά χώρα, πάντως η ποιότητα είναι πάντοτε το σημαντικότερο κριτήριο όταν θέλουμε να κρίνουμε προγράμματα και έργα και όχι ο αριθμός των ε, συμμετεχόντων. Τέλος, ε, συμφωνώ με τον Χάνου Τάκουλα και πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίζουμε προγράμματα και έργα που βασίζονται στην πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα και τα έργα. Και θα πρέπει τα κονδύλια να τα χρησιμοποιούμε έτσι, ώστε να επικεντρωνόμαστε στην πληροφόρηση ενημέρωση και μάλιστα στη γλώσσα των συμμετεχόντων. Χρειαζόμαστε επαφές στην εποχή της κρίσης και να μπορούμε να διασώσουμε ό,τι μπορεί ακόμη να διασωθεί. Πολύ ωραία και θαραλέα. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Α, όχι, ο κύριος Βάλγου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια φράση μόνο να πω. Κατάλαβα ότι στους διαγωνισμούς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική ισορροπία. Αυτό το θεωρεί σημαντικό η Κομισιόν. Δεν θα πρέπει όμως να δούμε μόνο γεωγραφικά το θέμα, αλλά τα ε, λιγότερο δραστήρια κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηριχθούν αυτά περισσότερο. Και αυτό πρέπει να ε, αντικατοπτρίζεται και στα κριτήρια για τους διαγωνισμούς. Ναι, Βέβαια, ε, τα χρήματα θα τα δίνουμε από την άλλη πλευρά σε αυτούς που προσπαθούν να τα ε, κατακτήσουν και να είναι άξιοι γι' αυτό. Ε, είναι λίγο μια προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου αυτό που ε, λέτε κύριε Μπάλκο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη και δεν θα θίξω το θέμα της νομικής βάσης αυτή τη στιγμή. Είμαστε ευτυχείς και καλωσορίζουμε στην Κομισιόν το γεγονό ότι η Επιτροπή σας ε, τώρα ε, μπαίνει στην ανάλυση της ίδιας της πρότασης. Ε, όπως υπόθηκε για τον εισηγητή, Υπάρχει πλέον μια γενικευμένη προσέγγιση από βράση του Συμβουλίου, η οποία φαίνεται να είναι ομόφωνη και αυτό ήταν και ένα από τα ζητήματα που ετέθησαν, δηλαδή αν υπήρξε κάποια αλλαγή ουσίας ανάμεσα στην πρόταση της Επιτροπής και την πρόταση που ενέκρινε το Συμβούλιο. Όχι, δεν υπήρξαν αλλαγές ουσίας. Μπορώ, ουσίας. Μπορώ να σας το διασφαλίσω αυτό και να σας καθησυχάσω. Υπήρξαν κάποιες μικρές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν μάλλον έτσι ένα χτένισμα του κειμένου ε, και επίσης ε, οργανώθηκαν λίγο καλύτερα τα στοιχεία που αφορούν ε, την οργάνωση και κάποια έτσι τυπικά στοιχεία. Επίσης ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ε, υπογραμμιστεί περισσότερο στο κείμενο του Συμβουλίου σε σχέση με αυτό που πρότεινε η Κομισιόν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν πραγματικά ουσιώδεις ε, αλλαγές. Επίσης, όταν μιλάμε για, αναφερόμαστε σε αυτούς που μπορούν να υποβάλουν έτοιμα για grants, το Συμβούλιο εδώ διήβρινε αυτό το πεδίο στις, ε, και συμπεριλαμβάνει πλέον και περιφερειακές αρχές, περιφερειακές οργανώσεις, καθώς επίσης και οργανώσεις, ε, πολιτιστικές οργανώσεις νέων. Επίσης, ε, κάποιες διατυπώσεις έχουν αλλάξει to όσον αφορά τις δέσμες και τις ε, κατευθύνσεις ε, ε, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και τα εγκλήματα τα οποία έλαβαν χώρα υπό απολυταρχικά καθεστώτα. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα τα οποία είναι, έτσι, αφορούν περισσότερο ουσιώδεις αλλαγές για όσον αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Συμφωνώ με τον εισηγητή και με άλλους ομιλητές ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα το οποίο έχει εκτιμηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ε, το νέο πρόγραμμα βασίζεται στις ε, επιτυχίες ε, του υφιστάμενου προγράμματος και οι διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και με τους δικαιούχους έχουν αποτελέσει μια πολύ καλή βάση μέχρι τώρα. Ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα πρόγραμμα bottom-up, διότι πράγματι βασίζεται σε σε, ε, ε, βασίζεται σε μια προσέγγιση βάσει της οποίας δίνονται τα grants σε αυτούς στους οποίους, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ε, και επομένως αυτή είναι μια καλή προσέγγιση κατά την απόψή μας και δεν πρόκειται να αλλάξει άλλωστε. Γνωρίζω ότι ε, προβληματίζεστε όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή. Είναι άλλωστε ένα μέλημα το οποίο ε, ανησυχεί και την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Θέλουμε να δούμε μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να διασφαλίσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και ισοτιμία, ισορροπία κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχουμε προτείνει ποσοστώσεις γιατί τέθη ένα ερώτημα επ' αυτού. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να, μέσα από άλλους τρόπους και με άλλα μέσα να επιτύχουμε την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή κυρίως μέσω της ενδυνάμωσης, της ε, ευαισθητοποίησης και της ε, γνώσης, ε, ειδικά στις περιφέρειες που μέχρι τώρα είχαμε μάλλον ε, χαμηλότερη συμμετοχή. Συμφωνώ απολύτως ότι αυτά τα προγράμματα δεν είναι μεγάλα, δεν είναι μεγάλο πρόγραμμα σε σχέση με άλλα προγράμματα και σίγουρα δεν θα είναι ελιτίστικο πρόγραμμα δεν έχουμε καθορίσει ποσοστά της 100. Ε, είπαμε ότι δεν μετράει το μέγεθος, αλλά η ποιότητα, καθώς επίσης και η επίπτωση των ε, προγραμμάτων. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία, αυτά μετράνε. Και βεβαίως κυρίως ε, η ποιότητα είναι το κύριο στατικό και το πιο σημαντικό για τέτοια προγράμματα σε γενικές γραμμές ε, πρέπει να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί τα πράγματα προχωρούν και προσδοκούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τη θέση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ε, και πραγματικά να σας καθησικάσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της έτσι ώστε να βοηθήσει την κατάσταση και έτσι ώστε να μπορέσουν να απαντηθούν τα διάφορα ζητήματα και να ενσωματωθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμείς ε, θέλουμε πάρα πολύ τα μεγάλα δίκτυα, μεγάλες NGOs, ΜΚΟ, να χρηματοδοτούνται και στο μέλλον. Όχι να ε, πρέπει κάθε φορά να ζητούν υποβολή προτάσεων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να καταστρέφουμε και ότι υπάρχει και να τα κάνουμε καινούρια οι υφιστάμενες δομές, τα δίκτυα που έχουν καταξιωθεί πρέπει να υποστηριχθούν για να συνεχίσουν να δουλεύουν γιατί λειτουργούν περισσότερο και για μακρότερο χρονικό διάστημα με επιτυχίες που τις επενέσατε κι εσείς ε, για μακρότερο χρονικό διάστημα από αυτούς, αυτά τα στελέχη της Κομισιόν που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Σύμφωνα με τον συνάδελφο Χάνου Τάκουλα ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η Κομισιόν από το μικρό προϋπολογισμό θα ε, καλύψει και την επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι ένα κομμάτι, αλλά η συνεργασία με τους πολίτες είναι κάτι διαφορετικό. Ο κύριος ε, Ρέπο, ο σκιώδης εισηγητής για τους σοσιαλδημοκράτες, ε, μην κάνετε ερωτήσεις ε, τώρα στην Επιτροπή. Θα, το, θα γίνουν από κοινού οι ερωτήσεις. Εμείς θα τις... Ε, ε, αποφασίσουμε. Γιατί έχω ακούσει ότι πολλοί απευθύνουν μετά ε, πιστολές στην Κομισιόν και με ερωτήματα. Θέλω να φανώ μια φορά και εγώ ευγενής προς την Κομισιόν και να τονίσω ότι εδώ είναι η ώρα που όλοι θα συζητούμε και θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Και αργότερα θα δουλέψουν οι σκιώδεις. Ευχαριστούμε Χάνου, καλή επιτυχία για το μέλλον και εύχομαι το Συμβούλιο και η Κομισιόν να ενδιαφερθούν για την έγκαιρη έναρξη του προγράμματος, γιατί παίρνω κάτι αγανακτισμένα σε επιστολές που λένε παρακαλώ μην επιτρέψετε να αποτύχει το πρόγραμμα. Βέβαια η Κομισιόν είπε ότι θα πρέπει να κινητοποιηθείτε τώρα, αλλιώς δεν θα έχει το 2014 πρόγραμμα. Όχι, θα πρέπει να έχουμε ε, ε, πρόγραμμα και αν δεν μας ακούνε, ε, δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, προχωρούμε στο επόμενο θέμα πριν από τους Ολυμπιακούς, ένα θέμα ενδιαφέρον η Διεθνής Αμνηστία για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στην Ουκρανία είδατε κάποιες συζητήσεις που δεν ήταν πάντα πολύ γόνιμες. Κάποιοι συνάδελφοι δεν πήγανε, άλλοι πήγανε και φρόντισαν για τη διαφάνεια, αλλά γενικά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της προετοιμασίας έπαιξαν ρόλο σημαντικό. Χαίρομαι που με προσήγησε η Διεθνής Αμνηστία και ανταποκρίθηκα αμέσω κι εγώ. Και χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Φράγκενταλ και η συνάδελφος από την Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, η κυρία Λόχ Μπίλερ. Μην χάνουμε χρόνο κύριε Φράγκενταλ, έχετε αμέσως το λόγο για 10 λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και σε εσά και σε όλου του βουλευτέ. Μα δίνει ευκαιρία τώρα να μοιραστούμε τι σκέψει μα όσον αφορά τον ε, ρόλο του αθλητισμού και όσον αφορά την δικιά μου για να κάνουμε να προσπαθήσουμε για να δούμε το συνολικό τοπίο. Θα δούμε ότι στον κόσμο σήμερα ο αθλητισμό έχει κατησχίσει τη πολιτική και ίσω και τη μουσική και τη τέχνη, διότι μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο, μπορεί να τον εμπλέξει, μπορεί να τονώσει τη φαντασία, να προκαλέσει συναισθήματα και να συνενώσει τον κόσμο και πολλές φορές βέβαια και να διχάσει. Ε, πρόκειται για κάτι το οποίο είναι παγκόσμιο, είναι κάτι πάνω από κουλτούρες, πολιτισμούς και εποχές. Και οι ήρωες του αθλητισμού έχουν γίνει δάλματα στην κοινωνία. Και οι βασικές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελο και η Ολυμπιακή είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτισμού και κουλτούρας. Έχουν γίνει κάτι σαν μαγνήτες για τα ΜΜΕ, για, τις για τα βασικά σήματα, μάρκες, για τους ε, χορηγούς, για τους εγκληματίες και όλοι αυτοί ελκύονται από τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τον αθλητισμό. Πρόκειται για ένα status symbol, ε, για τα χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις. Είναι κάτι που προκαλεί εθνικό καμάρι, περηφάνεια, να δεις κανείς τα επιτεύγματά του, να ελκύσει του, τουρίστες, ελκύσεις και πολλές φορές να κρύψει κάποια προβλήματα ε, τα οποία έχει με συγκεκριμένο κράτος. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τις εθνικές εκδηλώσεις μπορούμε να έχουμε μια, ε, μια, μια ενέργεια, μια, μια συμβολή καταλητική, να η, θετική. Γιατί πολλές φορές έχουμε να κάνουμε άμεσα με παραβιάσεις των Η ιδινή Αμνηστία έχει καταγράψει ε, επικοινωνίες εργασίας, ε, κατά τη διάρκεια των κατασκευών για κάποια εκδήλωση καταστολή των βασικών ελευθεριών όπως η ελευθερία του λόγου Αν την μεριά μπορεί να βοηθήσουν στην εξάπλωση και την, την ε, μία απεμπόληση των δικαιωμάτων όπως το λέει ο ΙΕ στο ψήφισμα του Οκτωβρίου 2011. Θα ήταν επομένω κάτι το πάρα πολύ δυνατό, σημαντικό, εάν δεν μπορούσαμε να ευθυγραμμίσουν τα δικαιώματα με τις αξίες, με τα, τα πρότυπα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Γιατί μπορεί ο αθλητισμός κάποιο είδους στερεότυπα που φέρνουν τις διακρίσεις να τα διαλύσει. Μπορεί να προωθήσει θετική εικόνα για κάποιους περιφερειασμένους. Ας πούμε οι παραολυμπιακοί πρόβαλαν ε, θετικές εικόνες για τους ε, αναπήρους και οι προσωπικότητες του αθλητισμού έχουν ε, γίνει διάσημοι και έχουν αλλάξει απόψεις και νοοτροπίες στον κόσμο. Ε, ο Τζεσι Όβενς, ο Μουχάμε Τάλι, Μπίλι Τζιν Κίνγκ, η Μαρτία Ναυρατήλοβα, η Βόμ Γκουλαγκόν, η Κάφια Φρίμα, ο Μπούλ Μπουλμερκά και άλλοι που έχουν συμβάλει ούτως ώστε να γίνουν ε, βήματα πρόοδου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διαφορετικούς τομείς και αναγνωρίζει την εισαπληνιστία τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο αθλητισμό όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αλλά το προβληματισμό μας αφορά σε πραγματικέ επιπτώσεις των βασικών ε, ε, εκδηλώσεων ε, εκεί που γίνονται κάποιες, κάποια, διοργανώσεις. Και αυτό ξεκινά στις κατασκευές όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και μετά γίνονται και κομμάτι της κληρονομιάς που αφήνουν οι οργανώσεις και καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτικών δικαιωμάτων, των ε, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία έκφραση, κίνηση, διακίνηση, συνεταιρίζεστε, ε, ελευθερία από ορισμένε διακρίσει, το δικαίωμα στην υγεία και στη στέγαση, είναι από τα βασικά δικαιώματα τα οποία ε, έχουν γνωρίσει παραδιάσει στα πλαίσια και εξαιτία διοργανώσεων. α πούμε, είχαμε πάρα πολλέ ε, εξώσει, αυθαίρετε ε, συλλήψει και παρενόχληση ε, αστέγων και μεταναστών κατά το παγκόσμιο κύπρο της Νοτιοαφρικής του 2010. Σε κάποιες χώρες πολλές φορές γίνεται χειρότερη η δεσμενή διάκριση κατά των γυναικών και πολλές φορές προσπαθούν οι οι αθλητικοί φορείς να εξασφαλίσουν, να να, να, να σιγουρέψουν την μη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό. Χρειάζονται επομένω κάποιο είδου επίγοντα μέτρα, ώστε να σταματήσει με αυτέ οι αρνητικέ επιπτώσει. Υπάρχουν κάποιε κυβερνήσει που δεν εξασφαλίζουν ε, τη, ζωή των δικαιωμάτων, θα πρέπει να κάτσουν στο εδόλιο. Και έχουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να λάβουμε κάποια μέτρα. να συμβουλεύσουμε δηλαδή, τα κρατημέλη όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει τόσο ώστε να μην συμβάλλει, τα μην συμβάλλουν στις καταχρήσεις των δικαιωμάτων και ούτως ώστε οι τρίτοι και αυτοί να έχουν πολλές λογοδοσίες. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε με κάποιους φορείς ε, αυτών των ε, διοργανώσεων, τόσο ώστε να έχουμε κάποια ελάχιστα στάντα, ελάχιστα πρότυπα και αυτά να τα εφαρμόζουμε. Επίσης θα πρέπει οι καλύτερες πρακτικές να λαμβάνονται υπόψη και να παρακολουθούμε το τι γίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τις οργανώσεις. Ε, βέβαια, συνήθως οι τρίτες χώρες ε, θεωρούμε ότι κάνουν τα πάνε σε αυτό το μέτωπο ε, και λέμε ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή δεν έχουμε πρόβλημα. Όμω από την άλλη μεριά, υπόψη τι γίνεται σε διάφορε διοργανώσει και στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου που μας οδηγούν σε αντίθετο συμπέρασμα γιατί έχουμε τρία θέματα που αξίζουν προσοχή σε σχέση με τους Ολυμπιακούς του 2012. Πρώτα πρώτα τα δικαιώματα των εργαζομένων τα παρέβησαν οι κλάδοι των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων. Επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με το τι κάνανε οι χορηγοί και επίση η βία των γυναικών. Σύμφωνα με κάποια έκθεση με οργανώσεων και ε, συνδικάτων, με ένα φορέα που ονομάζεται Playfair, οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατασκευάζουν ε, κάποιε πάρα πολύ προβλημένε μάρκε και ε, κεντρικά καταστήματα πληρώνονται πάρα πολύ χαμηλού μισθού, του ζητάνε να δουλέψουν ε, με τρομερέ υπερορίε και του απειλούν με απόλυση. επισκέφθηκαν. Οκτώ εργοστάσια με αγαθά και στους στου σε Κίνα, Φιλιππίνη και Σιλάνκα και είδαν ότι υπάρχουν πάρα πολλέ παραβιάσει των δικαιωμάτων και αυτό τα γράφει η έκθεση που συνετάγει. Οπότε, λόγω αυτής της έκθεσης της Playfair, ε, η Ολυμπιακή Επιτροπή για το Λονδίνο απίτησε να γίνει συμμόρφωση λοιπόν και να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί καταγγελία, ούτω ώστε να, υπάρχει, να υπάρχουν καταγγελίε, να υπάρχει έρευνα, να υπάρχει αποκατάσταση των παραβιάσεων. Επίση είπαμε ότι θα πρέπει και κάποιοι αμερόληπτοι να φτιάξουν κώδικα διοντολογία και αυτό να εφαρμοστεί στου ολυμπιακού του Ρίο σε τέσσερα χρόνια. Πολύ βασικό αυτό. Ε, κάτι άλλο που γίνεται στι μεγάλε εκδηλώσει αφορά τους ε, χορηγούς και τις συστάσεις τους υπήρχαν που έχουν γιατί αυτό το εξετάσαμε πάρα πολύ αυστηρά σε σχέση με, το 2012. Θα θυμάστε τι έγινε το 1984 στον Ποπάρα στην Ινδία που είχαμε κάποια τοξικές διαρροές και εδώ πέρα ε, πρόκειται για μια περίπτωση βαριτά της αμήλης ο λόγω καυστερίας και ε, τελικά έτσι εφήγησαν ε, τα δικαιώματα στην υγεία, στην ίδρυυση, στην, ε, στο επίπεδο διαβίωση, ε, τα δικαιώματα που 100.000 άτομα. Και από το 2001 η εταιρεία χημικών Dow είναι ο μόνος ε, κύριος της εταιρείας Γιώργη Καρβάλη. Το 1910 τον Ιούνιο η Dow έγινε Ολυμπιακός εταίρο και τον Αύγουστο του 2011 ε, είδα μια μεγάλη δουλειά σε αυτό το Ολυμπιακό στάδιο και αυτό προκάλεσε αγανάκτηση μεγάλη στην Ινδία. Και σε υπουργικό επίπεδο γίνανε καταγγελίε. Η Ολυμπιακή Επιτροπή τη Ινδία ε, ε, ε, ενεκάλεσε την ε, Ολυμπιακή Επιτροπή για το Βενδίνο. Αλλά δεν έκανε πίσω η Ολυμπιακή Επιτροπή και αυτό σημαίνει ότι για τη σύμβαση δεν λήφθη υπόψη η περιοχή τη εταιρεία Ντάου στο παρελθόν. ακόμα εκκρεμούν ε, καταγγελίες για αποζημίωση, για επανόρθωση, για το πώς η ΝΤΑΟ θα βοηθήσει τους επιβιώσαντες ε, σε σχέση με την πρόσβαση σε νερό κλπ. Επίση, είναι πάρα πολύ βασικό το θέμα της βίας κατά των γυναικών, της βία κατοίκων, σεξουαλική βία, ε, δουλεμπορία γυναικών, εκπόρνευση και πολλές φορές αυτοί που είναι από το περιβάλλον των γυναικών αθλητριών και αυτοί, ε, και αυτοί τους κακομεταχειρίζονται. Πολλές φορές αυξάνεται λοιπόν η πορνεία ε, κατά τις διοργανώσεις, οπότε έχουμε πιο πολλές γυναίκες που είναι αντικείμενα ε, εκπόρνευσης και άλλων ε, κακοποίησεων σεξουαλικών. Και επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είχαμε διπλασιασμό των, ε, της δραστηριότητας της ε, εμπορίας ε, ανθρώπων και γυναικών επίσης για και είδαμε ότι μετά δεν έπεσε, μετά τους δεν έπεσε αυτός ο δείκτης Επομένω είναι πάρα πολύ βασικό το πώς κατά αυτά τα γεγονότα οι οργανωτές, η αστυνομία, ε, η κυβέρνηση και κυρίως οι γυναικοί φορεί να συνεργάζονται, ούτω ώστε να μπορούν να υπολογίσουν τι κίνδυνοι υπάρχουν και να μπορούν να έχουν κάποια ε, μέτρα πρόληψης. Ε, και αυτό να γίνεται πολύ νωρίτερα του αθλητικού γεγονότος. Και δεν μας εξέπληξε το ότι οι διεθνεί ομοσπονδίε όπω η FIFA και η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή κάνουν πάρα πολύ λίγο όσον αφορά το πώ θα προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλούμε τώρα για διεθνικού φορεί, ε, μη κυβερνητικού, που θα πρέπει αυτού του οργανισμού, αυτού του φορεί να του πιέσουμε να σεβαστούν τα δικαιώματα. Η Ολυμπιακή Επιτροπή θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. σε συνεργασία με τι Εθνικέ Ολυμπιακέ Επιτροπέ. Έτσι θα αφήνουμε περισσότερο αυτά που θέλουμε και επίση ε, με την FIFA θα μπορούσε να απαιτήσει από τα μέλη να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί κατά την φάση των προτάσεων και όλοι όσοι ζητούν να φιλοξενήσουν κάποιε διοργανώσει, θα πρέπει να υποβάλουν προγράμματα ενδελεχή για το πώς θα συμπροσθέσουν τα δικαιώματα και επομένω, ε, η μελέτη αυτή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική και απαραίτητη. το, το, το, το τελικό, τελευταίο ερώτημα είναι το εξή. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι αρμοδιότητέ τη, σε σχέση με την ε, πολιτική που έχει κηρύξει για αυτέ τι αρνητικέ διοργανώσει και πάντα στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά το στρατηγικό πλαίσιο το οποίο θεσπίστηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να δεσμευτεί όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων, όσον αφορά το να εντάξει την πόλη των δικαιωμάτων στην νέα πολιτική αθλητισμών. θα πρέπει να επεξεργαστεί ε, με ένα σχέδιο τόσο ώστε ε, να εξασφαλίσει την τήρηση αυτού του πλαισίου που συζητούμε την σε σχέση με τι υποχρεώσει τη των κρατών μελών. Να εξασφαλίσει την τήρηση και όποτε χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με κάποια κοινά πρότυπα να εξασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και σε σχέση με τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καλύψει κάποια προγράμματα για προστασία των δικαιωμάτων και για το mainstream και την ένταξη τη πολιτική των δικαιωμάτων. Το 2011 η Επίτροπος Βασιλείου επισκέφθηκε ε, την έδρα του ε, Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λοζάνη και ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια του διαλόγου άρχισε τότε μεταξύ Επιτροπή και Ολυμπιακού Κινήματο ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει μόνο για εκείνη την, την, εκείνο το διάστημα, ώστε να, πιώσει, να πιέσει, συγγνώμη, να πιέσει, ούτω ώστε να ισχύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά τη διαδικασία τη επιλογή και για, το, για, τα, για, από τους προμηθευτές και από τους χορηγούς. Για Ολυμπιακούς Αγώνες και αζαδικές εκδηλώσεις. Το Κοινοβούλιο τώρα. Εμείς να έγκληση στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δεσμευτεί απολύτω όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων στα πλαίσια αθλητικών εκδηλώσεων. Και θα ε, εκφέρουμε έκθεση στο Κοινοβούλιο να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να συγκροτήσει ό,τι οι πολιτικέ χρειάζονται και οτιδήποτε ρυθμιστικά διαδήματα να αναλάβει, ούτω ώστε να αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλήσει η Επιτροπή σα σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή του Ανθρώπινου θα μπορεί να παρακολουθεί και να πρέπει να παρακολουθεί τι γίνεται με τα δικαιώματα στις, και τι επιπτώσεις υπάρχουν. Και επίσης θα πρέπει να αναφέρει σχετικώς στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει τα, οι οργανώσεις, οι αθλητικές, να αποτελούν υπόδειγμα σεβασμού των δικαιωμάτων. Και για να προσέξουμε λοιπόν σε όλε τι πτυχέ του προβλήματο, χρηματοδότηση, διαχείριση, θέση εμπορία, έχουμε μακρύτερα μπροστά μα και επομένω νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαμετρήσει σημαντικό ρόλο σε πρόθεση αυτού του οράματο και θα χρησιμοποιήσει τι ε, αρμόδιε αυτέ, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα θα είναι ένα πρόσωπο τμήμα τη προσέγγιση που έχουμε για τι θετικέ εκδηλώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυρία Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την αμνηστία για την πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση. Αρχίζω με τα θετικά, γιατί νομίζω ότι πριν από λίγα χρόνια θα θυμούνται μερικοί από εμά το 1978 με την ε, δικτατορία στην Αργεντινή. Κανένας ε, Ευρωπαίος πολιτικός δεν το είπε θα είχαμε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου εκεί και λίγοι μίλησαν γι' αυτό στην Ευρώπη. Τώρα έχουμε πολλές ευκαιρίες όπου συνηθίζεται πολιτικοί να μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες όπου είναι κακή η κατάσταση Και λίγες είναι οι διοργανώσεις οι αθλητικές εκεί. Το είπατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε στην αρχή με το ποδόσφαιρο στην Ουκρανία το πρωτάθλημα, είχαμε του Άσ Χόκκι στη Λευκορωσία, ε, στο Σότσι η χειμερινή ε, Ολυμπιακή, παρά τη σοβαρή καταπίεση των ανθρώπων εκεί. Οπότε είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε όλες τις σφαίρες της πολιτικής. Λίγα θα προσθέσω στην παρουσίαση της Διεθνούς Αμνηστίας. Από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να δούμε και τα δικαιώματα των ίδιων των αθλητών. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα αν σε κάποιες χώρες οι αθλητές αναγκάζονται να παίρνουν φάρμακα και να το πάρονται για να έχουν επιδόσεις υψηλές. Και το κάνουν αυτό καμιά φορά χωρίς να έχουν γνώση και χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι αθλητές πολλές φορές μπορεί να είναι ε, πρεσβευτές ε, ειρήνης, ε, καταλήτες, το είδαμε αυτό ήδη. Άνθρωποι δραστήριοι εντάχθηκαν σε επαγγελματικές ομάδες και έπαιξαν με αντιπάλους τους για την αλλαγή. Επίσης ο χάρτης τη Διεθνού Ολυμπιακής Επιτροπή λέει ότι ο αθλητισμός είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Όλοι συμφωνούμε. Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ε, ασχοληθεί με το σπο, με τον αθλητισμό, χωρίς διακρίσεις, στο, με το ολυμπιακό πνεύμα, αμοιβαία κατανόηση, φιλία, αλληλεγγύη, εφαγωνίζεστε. Δεν ακούγονται μόνο καλά, είναι καλά αυτά. Και αν δούμε τις πρακτικές των διαφόρων χωρών βλέπουμε ότι υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάσεις των πρακτικών. Δείτε τη Σαουδική Αραβία όπου τα κορίτσια δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ε, τάξεις γυμναστικής ε, και οι γυναίκες και τα κορίτσια απαγορεύεται να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς. Εδώ υπάρχει σαφής παραβίαση της σύμβασης του ΟΗΕ ε, κατά των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Παραβιάζει η Σαουδική Αραβία και αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας στην Επιτροπή μας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δικαίωμα άσκησης του αθλητισμού είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Φράγκενταλ από την Αμνηστία αναφέρθηκε ήδη στη μεγάλη ευθύνη των αθλητικών ε, οργανώσεων ε, όπως FIFA κλπ. Αυτές οι οργανώσεις θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ακριβείς και συγκεκριμένες όταν μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, επιταγές που απορρέουν από αυτές. Όταν μιλάμε για την Κίνα και τους Ολυμπιακούς, όταν απευθύνονται στην κοινή γνώμη, λέει ναι, συμφωνήσαμε να βελτιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά επί χάρτου δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μια προφορική δήλωση μόνο του αντιδημάρχου του Πεκίνου. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι όταν διαπραγματεύονται και αποφασίζουν σε ποιους θα αναθέσουν τους Ολυμπιακούς. Αλλά υπάρχουν και άλλες αθλητικές ε, οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο που είναι πολύ σημαντικές για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη χώρα μου, τη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε μια ομοσπονδία, την Γερμανική ε, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπου ε, έχουν μέλη η γερμανική δηλαδή ε, ποδοσφαιρική έτος έχει περίπου 7 εκατομμύρια μέλη και 26.000 λέσχες ε, ζηλεύουν τα πολιτικά κόμματα. Έχουν μια δομή λοιπόν ε, που αν τη χρησιμοποιήσουν για να πειράσουν τους νέους και τους ενήλικες επίσης θετικά θα πετύχουν πολλά κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων. Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πριν από λίγο καιρό υιοθέτησε ένα θετικό πρόγραμμα ε, για τα μέλη τους για να τα εκπαιδεύσουν κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού που έχει τόσο φρικτά αποτελέσματα όπου χαιρετίζουν χιτλερικά πολλές φορές και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές ε, που όταν δεν είναι λευκοί αντιμετωπίζουν μεγάλη βία και επιθετικότητα και η Επιτροπή σας λοιπόν θα μπορούσε να συζητήσει με άλλες αθλητικές ε, οργανώσεις και ομοσπονδίες ώστε αυτές να ασχολούνται περισσότερο μόνιμα με τα θέματα αυτά. Επίσης από τα Συμβούλια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε το ψήφισμα του 2010 που λέει συγκεκριμένα ότι η μάχη κατά του ρατσισμού είναι πολύ σημαντική και πρέπει να απασχολήσει και τις αθλητικές ομοσπονδίες. Αυτά που είπατε κυρία Φράγκενταλ σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, τα σημείωσα, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Επίσης έχουμε μία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας και τις εταιρείες όπως Union Carbide στο Βοπάλ. Υπάρχουν και άλλες όπως η Adidas και η Puma που φτιάχνουν αθλητικά είδη και θα μπορούσαμε να τις ενθαρρύνουμε περισσότερο να έχουν ε, περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες να συμμετέχουν στο δίκαιο εμπόριο κλπ. Και εγώ να προσθέσω κάτι το οποίο ε, ε, σημείωσα και στην έκθεση φύσας που κατέθεσα και τροπολογία. Ε, είχαμε μιλήσει για τις ε, διακρίσεις σε βάρος των γυναικών ε, πριν από τους Ολυμπιακούς στην Αγγλία και μου είπαν ότι το πρόβλημα είναι ότι όλο και οι περισσότερες γυναίκες επειδή δεν αναγκάζονται να ακολουθήσουν ε, τις αυστηρές επιταγές του Ιράν. μια φορά στο Ιράν έπαιξε η γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα και είχε ντυθεί όπως δίνονταν οι γυναίκες στο Ιράν. Αν πάμε σε αυτό το επίπεδο δεν εκπλήσει ότι μετά όλα αυτά βρίσκουν μιμητές. Και επίσης στο Λονδίνο οι κυρίες μου είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Παλιά ήταν καλύτερα τα πράγματα και τώρα χειροτερεύουν γιατί εμείς οι δυτικοί θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, τους προσεγγίσουμε, τους Ιρανούς ας πούμε, και να αντιθούμε και εμείς όπως συντείνονται οι Ιρανές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και για τους ε, Ολυμπιακούς Αγώνες. Και η Ολυμπιακή Επιτροπή, αν βασιστεί στο χάρτη της, ε, θα το καταπολεμήσει αυτό το πράγμα. Υπάρχει σαφής ε, πρόβλεψη για αυτά τα πράγματα στην, στον Ολυμπιακό χάρτη. Πολλές φορές επιμένουμε στα πολιτικά ορθό ή όχι, αλλά ο κώδικας ενδυμασίας ε, πρέπει να είναι δεδομένος και να τηρείται. Και αν βλέπω ότι οι Γερμανοί ε, όταν ε, οι Γερμανίδες όταν έπαιζαν στο Ιράν, μιμούντο τις γυναίκες στο Ιράν, πρέπει να πω ότι αυτό δεν βοηθάει τις γυναίκες στο Ιράν οι υπεύθυνοι λοιπόν για τον αθλητισμό, για τις μεγάλες διοργανώσεις θα πρέπει με μεγάλη αυστηρότητα να επιμείνουν να εφαρμόζεται ο χάρτης και οι κανόνες που πρέπει να ισχύουν για όλους και δυστυχώς δεν ισχύουν. Τώρα ο κύριος Μπόρις, ο κύριος Κουρία και μετά ο κύριος Μιγκάλσκι. Κύριε Μπόρις. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μόλι τώρα τέλειωσε το γύρο στην Πολωνία, κατά τη γνώμη μου. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ήταν επιτυχή αυτή η εκδήλωση, αλλά και τα πήγαμε καλά για αυτό το οποίο μας απασχολεί τώρα. Ξέρετε, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να αλλάξουμε κάποια στερεότυπα. Το ίδιο ισχύει νομίζω για το Παγκόσμιο Βιβλίο τη Αφρική. Ο κόσμο έτσι μπόρεσε έτσι να ανακαλύψει αξίε που δεν ήξερε, έτσι μπόρεσε να επιδείξουμε ελεγγύη και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνονται θαραλέε αποφάσει όσον αφορά ε, τέτοιου είδου διοργανώσει και γι' αυτό επίση να δούμε πόσο ε, όλα αυτά είναι σημαντικά σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. επίση να είδατε τι έγινε και με τους ε, Ιταλού που έπαιζαν στην χώρα μας. Τι έγινε επίσης... Ε, ε Όπω έγινε με τον Παλατέλη που παίζει στην Ιταλία που είναι μαύρο, που έγινε και με ένα δικό μα που είναι μαύρο και παίζει για την ομάδα μα. Καλύτερη ευκαιρία είχαμε να αναδείξουμε ε, αυτό το, το, στερεότυπο, το καινούριο, σε σχέση με, τις, με τα παιχνίδια σε εθνικό επίπεδο. Όλοι αυτοί γίνανε εθνικοί ήρωε ε, με, με τα επιτυχία αποτελέσματα. Γι' αυτό και νομίζω ότι η συμμετοχή αυτών των μαύρων παικτών στην, ε, στην εθνική ομάδα ε, πιάνει τόπο περισσότερο από το να εξοδεύει ε, εκατομμύρια σε ενημερωτικέ εκστρατείε. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο αθλητισμό μπορεί να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό, μπορεί να καταπολεμήσει τι νέε διακρίσει Να μερικά αποτελέσματα αυτά, ε, μερικά παραδείγματα σαν γι' αυτά που αξίζει να τα σκεφτούμε, τα λάβουμε από πολιτική. πολιτικής. είδαμε τη ίσχυσε όσον αφορά την Ουκρανία, τη ίσχυσε όσον αφορά τις διαμαρτυρίες, τις εκδηλώσει κατά της παραβίασης των δημοκρατικών αρχών στην, ε, Ουκρανία. Κανείς δεν ε, καταφέρθηκε κατά ε, την αθλητικών εκδηλώσεων. Όμω κάποιοι πολιτικοί δεν πήγαν στου στους αγώνες στην Ουκρανία. Γιατί είπαν δεν θέλουν να πάνε σε κάποια χώρα που φέρεται έτσι ο πολιτικής Οπότε έτσι, έτσι τώρα ο κόσμο θα προβληματιστεί. Οι Ουκρανοί, και αν όχι η πολιτική, τουλάχιστον ο κόσμο, θα, θα κάνει διαφορετικέ επιλογέ και θα ψηφίσει αλλιώ. Είναι πολύ σημαντικό μέσα αυτό το οποίο έγινε. Γιατί έτσι μπορεί ο κόσμο σε μια χώρα να, να καταλάβει ότι η Ευρώπη κάποια πράγματα τα βλέπει αλλιώ όταν βρίσκεται στη χώρα του. Και επίση Και εγώ συμφωνώ ότι κάθε μεγαλύτερη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προσβασιμότητα των αναπήρων στα, στα παιχνίδια, στο, στα, στις αθλητικές συναντήσεις. Και έχουμε διάφορε μορφέ αναπηρία. Α πούμε, είχαμε ένα πρόγραμμα στη χώρα μα. Αυτό το πρόγραμμα Ε, αφορούσε το, το, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μια που δεν μπορούσαν να δουν οι τυφλοί, τους δώσαμε ακουστικά και επίσης ε, όντας μέσα στο στάδιο μπορούσαν να αισθανθούν την ατμόσφαιρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να γίνονται για κάποιες ομάδες ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες. Άρα αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Το πώς θα έχουμε αυξημένη προσβασιμότητα για τους, ε, για, τους αναπήρους. Ο κ. Ε, εγώ θεωρώ, αγαπητέ κύριε Δημοκυρμά που μιλάω από την πλάτη ότι ήταν πάρα πολύ αμήχανα σε σχέση με την διοργάνωση αυτή. Εγώ θεωρώ ότι είμαι σαν ένα. Πάρα πολύ σαν μεγάλη πίεση. Ενοχλούμε αυτό τον κύριο Καβαλέγκα που είναι πολιτικό κρατούμενο στην Λευκορωσία. Θα πρέπει επομένω να αναγνωριστεί ότι αυτός ο κύριος είναι ε, φυλακισμένος για λόγους ε, συνείδησης. Ε, απευθύνθηκα στις αρχές, πιθανόν σε επαφή μαζί του όμως ήταν αδύνατο, διότι είχαμε την πολιτοφυλακή οι οποίοι προέβησαν σε αυτήν την, τη σύλληψη. Τέλο πάντων ήταν τελείω θολό, τελείω ασαφέ το ποιο είχε δίκιο ή όχι. Τώρα, εν πάση ε, κρατείται στη φυλακή. Κάνει απεργία πείνα εδώ και δύο μήνε. Και κάθονται και μα λένε, λένε στην, στην, ε, στην Διεθνή Αμνηστία ότι αυτό φταίει γιατί αυτό έδειρε του αστυνομικού. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολλά η Διεθνή Αμνηστία και νομίζω ότι έχει καταφέρει να αποφυλακιστούν χιλιάδε. Χιλιάδε κρατουμένων και με την ευκαιρία ευχαριστώ για την κατανοησή σα. Και μας λέτε τώρα ότι η αμνηστία σε σχέση με τους Ολυμπιακούς ε, προσπαθεί να δει ποιος ωφελήθηκε πόσο, τι γίνεται όσον αφορά τα, τα οικολογικά πρότυπα. Αλλά προσέξτε μήπως, μήπως ο Ολύμπος στρέφεται προς αυτά και ξεχνάτε αυτός που είναι στη φυλακή τόσο καιρό. Σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχω τώρα Δύο ερωτήσει σε αυτό που συζητήσαμε. Έχουμε στη Λευκορωσία ε, διεθνείς αγώνες χόκι και επίσης άλλη μια διοργάνωση στο Σότσι. Μήπω η Διεθνή Αμνηστία πρέπει να απαιτήσει να αλλάξει ο τόπο διοργάνωσης ε, αυτών των αγώνων. Ήδη έχουμε πει ότι θα πρέπει το χόκε να μην γίνει στην ε, Λευκορωσία. Πρόκειται περί δικτατορίας. Δεν είναι το σωστό μέρος για τέτοια διοργάνωση. Αλλά και για τους Ολυμπιακούς του Σότσι, τους χειμερούς Ολυμπιακούς του Σότσι της Ρωσίας. Γιατί άλλωστε το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι ήταν ενώθες εκλογές που έγιναν τότε. Δεν είναι δυνατόν όμω έχουμε αυτέ τι δύο εκδηλώσει που να γίνουν σε αυτέ τι χώρε που έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν φυλακισμένοι για λόγου συνείδηση. Ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη ερώτηση στον κύριο Φράγκενταλ. Θα ήθελα να καταλάβω, λαμβάνοντα υπόψη και την επιρροή που έχει η οργάνωση Διεθνή Αμνηστία στην διεθνή κοινή γνώμη, παγκόσμια κοινή γνώμη, αλλά και σε πολλέ ε, κυβερνήσει εάν είχε γίνει κάτι όσον αφορά την ε, διακριτική μεταχείριση των γυναικών ε, στον αθλητισμό ε, σε ορισμένες Ισλαμικές χώρες. Να καταλάβω δηλαδή εάν ε, το γεγονός ότι τέτοιες γυναικείες ομάδες δεν συμμετέχουν στο ε, Λονδίνο, εάν ε, αποτέλεσε έτσι ξεκίνημα για δράση οποιαδήποτε, οποιοδήποτε είδους από τη Διεθνή Αμνηστία. Επίσης, στην Κίνα είχαμε ε, ε, θριαμβευτικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Επομένως θεωρώ ότι οποιαδήποτε περαιτέρω θεώρηση για άλλες περιοχές που λαμβάνουν χώρα Ολυμπιακοί Αγώνες περιτεύει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ναι, βέβαια δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα όπως θα, όπως θα έπρεπε. Είμαστε ένα κοινοβούλιο που δεν μπορεί να υπερβεί τις αρμοδιότητες του. Μπορούμε να εγκρίνουμε ψηφίσματα όμως που καμιά φορά τα ακούν, τα επικρίνουν, τα ακούν πολύ. Η Κίνα, για παράδειγμα, τα προσέχει πολύ και αντιδρά αλλεργικά στα ψηφίσματά μας. Αλλά και η Επίτροπος Βασιλείου και άλλοι θα μπορούσαν να παρέμβουν. Θα μπορούσαμε να απευθύνουμε εκκλήσει σε πολλούς, σε εκείνους που αναθέτουν τις διοργανώσεις ή εκείνους που είναι σε διάφορα εποπτικά όργανα ή εκεί όπου γίνονται κληρώσεις, ούτω ώστε να είναι ξεκάθαρο από την αρχή ότι χώρες ε, που, όπου υπάρχουν πολλές παραδιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν να συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν διοργανώσεις. Και αυτό πρέπει να παρουσιαστεί ως λόγος. Αν κάνουν όλοι πίσω και δεν τολμούν να πούν ότι ναι, γι' αυτό το λόγο, ίσως και για λόγους οικονομικούς, συνήθως οι οικονομικοί είναι οι λόγοι, δίκιο έχεις τότε περιοριζόμεθα. Δεν πρέπει να ζητάτε υπερβολικά πολλά πράγματα από εμά, αλλά μπορούμε να βάζουμε πάντα το δάχτυλο επί των τύπων, των ύλων και η Επιτροπή, Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, ε, κάνει μεγάλη προσπάθεια εδώ. Η Πέτρα. Όχι, τα πιο σημαντικά τα είπαμε ήδη. Είναι σημαντικό που είπατε σε ποια σημεία μπορούμε να κάνουμε κάτι, σε, ποια, ε, σε ποιες υπηρεσίες. Πάντως η βασική ευθύνη είναι στις ομοσπονδίες, στις αθλητικές ε, οργανώσεις. Συζητάμε για παράδειγμα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην, στην Ουκρανία σε μια περίοδο όπου υπάρχει μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ενώ γίνονται οι συζητήσεις αυτές, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπολ, ε, πάλι αναθέτει τη διοργάνωση στην Ουκρανία. Δηλαδή αναρωτιόμαστε, καταλαβαίνουν, φτάνουν οι συζητήσεις μας αυτές τις ομοσπονδίες, εκτός και αν πραγματικά πρόκειται μόνο για τα λεφτά. Πάντως πρέπει να ξεκαθαρίζουμε ξανά και ξανά στις ομοσπονδίες ότι ο αθλητισμός μπορεί να παίξει πολύ ενωτικό ρόλο, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι αποφάσεις που λαμβάνει για το πού θα γίνει μια διοργάνωση. Αν θα ανατεθεί σε μια χώρα μια διοργάνωση ή όχι. Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτεί κάποια πράγματα όταν συνοδεύεται από μια σωστή αιτιολόγηση που θα λέει όχι εκεί διότι υπάρχει μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουν πολιτική και κοινωνική ευθύνη και οι ομοσπονδίες. Ευχαριστώ. Να δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Φράγκενταλ ή ε, στην συνάδελφό του που ε, ήταν παλιά μου συνεργάτη στο γραφείο μου. Κύριε Φράγκενταλ, τι έχετε να παρατηρήσετε και να απαντήσετε σε αυτά που ακούσατε εδώ. Α, έδωσα το λόγο στον κύριο Φραγκεταλή. Κυρία Μπενεραπατού. Α, η κυρία Μπενεραπατού. Ναι, είχα ζητήσει το λόγο ήδη. Έχουμε λίγο την αίσθηση ε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μια αίσθηση αδυναμίας. Ε, και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στην κυρία, ε, στη συνάδελφό μας, αλλά και στον εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμυστίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κινητοποίηση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέτρεψε την αλλαγή προγράμματος ή την αποτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο πραγματικά στον κύριο Φράγκερ. Παρακαλώ. Many very... Ε, ε, θέθησαν πολλά ζητήματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά από αυτά. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι συμφωνώ μαζί σας κυρία Πρόεδρε ότι αυτό που μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μάλλον ε, περιορισμένο. Ε, μπορεί βεβαίως ε, να περάσει ψηφίσματα και να κάνει και τηλεφωνήματα προς διαφόρους ανθρώπους, να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη φήμη του και την πίεση του έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα και δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Σαφές ε, είναι ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, δυνατότητες και ευκαιρίες. Ο κύριος Μιγιάννης και αναφέρθηκε στα μεγάλα μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να λάβουν χώρα σε κάποιες ε, ε, χώρες. Κοιτάξτε, ε, πρόκειται για αμφιλεγόμενα ζητήματα. Η Διεθνής Αμνηστία δεν συμμετέχει σε μποϊκοτάρισμα τέτοιων διοργανώσεων. Ε, γιατί θα πούμε ας πούμε όχι σε μια διοργάνωση ε, στη Λευκορωσία και μετά θα αφήσουμε κάτι να γίνει στην, ε, στην Κίνα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαδικασία η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και άλλες μεγάλες αθλητικές οργανώσεις ε, έχουν κατά κανόνα στον ε, κανονισμό λειτουργία τους ε, και κεφάλαιο που αφορά την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από εκεί απορρέουν συγκεκριμένες ε, υποχρεώσεις. Επίσης ε, υπάρχουν στρατηγικά πλαίσια, ε, σχέδια δράσης, υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την κύρωση και υπογραφή διεθνών συμφωνιών κτλ. Τώρα, η κατάσταση στην οποία θέλουμε να φτάσουμε είναι οποιαδήποτε κυβέρνηση ε, οργανώσει κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός να ξέρει ότι οπωσδήποτε θα μελετηθεί ε, σε λεπτομέρεια το μητρό της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, παραβιάσεις. και ότι δεν θα αφήσουμε να περάσει ασχολίαστη οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και η FIFA και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ε, το γνωρίζουν αυτό. Ε, υπάρχουν και σχετικές οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά πρέπει να είναι σαφή μηνύματα έτσι ώστε να ξέρουν οι διοργανώτες χώρες τι τους περιμένει. Γιατί διαφορετικά θα βρεθούν σε δυσάρεστη θέση, σε άβολη θέση όταν θα είναι έτοιμες να διεκδικήσουν την την διοργάνωση την οποία θα διεκδικήσουν. και ε, να γνωρίζουν ε, επίσης οι χώρες ότι αν υποβάλουν υποψηφιότητα για ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός ε, θα μελετηθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά ε, την, ε, τις ε, γυναικείες ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και άλλες αραβικές χώρες, Εμμυράτα κτλ. Την, τον αποκλεισμό γυναικείων ομάδων. Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Και βεβαίως την στιγμή των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων βρίσκουμε την ευκαιρία ε, να συζητήσουμε θέματα σαν αυτό και αν η Σαουδική Αραβία θέλει πραγματικά να βρει τη θέση της στο διεθνές στερέωμα και το αθλητικό και το πολιτικό θα πρέπει να ξεπεράσει τέτοιου είδους ε, προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φράγκενταλ. Νομίζω ότι ήταν ε, χρήσιμο ε, να σας ακούσουμε αυτή τη ε, στιγμή. Μεσολάβησε η συνεργάτη σας και πραγματοποιήθηκε η συνάντησή μας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς προσπαθούμε να λαμβάνουμε υπόψη μας όσο γίνεται πιο συστηματικά. τουλάχιστον ενώπιον των οργανισμών που είναι υπεύθυνε για τα ζητήματα αυτά. Ε, θέλουμε πάντα να γίνεται αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε δύναμη από μόνοι μας Εμείς βέβαια έχουμε ε, τις ανευρωπαϊκές χώρες ε, και την Χάρτα των Θεμελιδών Δικαιωμάτων ε, και βεβαίως είναι πάρα πολύ καλό πολλές, πολλές οργανώσεις να προσυπογράφουν αυτά τα ιδεώδη της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να κάνετε και μια μικρή έκθεση πάνω σε αυτό. Γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι πάντα στην επικαιρότητα να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη λέγοντας, ε, αναφέροντας συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ε, σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες οργανώσεις, ε, συγγνώμη, σε συγκεκριμένες διοργανώσεις δεν έγινε σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι συγκεκριμένες αθλητικές οργανώσεις έδωσαν σε ορισμένες χώρες την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών ε, συμβάντων χωρίς να λάβουν υπόψη τον μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας. Και τώρα ολοκληρώνουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, πρέπει να φύγουν όλοι πλην των συντονιστών. Μην ξεχάσετε αύριο να φέρετε και τις κάρτες ψηφοφορίας σας παρακαλώ.